Uh, uh, Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας καλησπερίσω. Χαίρομαι ιδιαίτερα που υποδέχομαι τον Βίνσεν Βαν Κίκενμπόρν, ο οποίος είναι ο Βέλγος Υπουργός για τα θέματα απλούστευσης. Ε, πρώτη φορά το ακούμε, αλλά είναι κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Πριν του δώσω το λόγο. Θα ήθελα να κηρύξω την έναρξη επισήμως πλέον της ε, σημερινής μας συνεδρίασης. Έχετε μπροστά σας την ημερήσια διάταξη, το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Ε, σα ζητώ να το εγκρίνουμε. Και να σας πω ότι επίσης ε, ε, η συνάντησή μας υπόκειται σε web streaming. Δηλαδή, να ξέρετε ότι από τη στιγμή που πατάτε το κουμπάκι για να πάρετε το μικρόφωνο, η εικόνα σας θα εμφανίζεται στο διαδίκτυο. Είναι πραγματική, πραγματικά τιμή για, με, για μας, για όλους που είσαστε μαζί μας στην αρχή της Βελγικής Προεδρίας για να ακούσουμε από τον Υπουργό, τον Βίσεν τα θέματα εσωτερικής αγοράς. Εάν δείτε και το έγγραφο το οποίο διανεμήθηκε, η εσωτερική αγορά και η ανταγωνιστικότητα είναι ένα από τα θέματα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Βελγική Προεδρία. Λοιπόν, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Υπουργό για να μας μιλήσει για κάποια αυτά τα θέματα. Επίσης, η Βελγική Προεδρία έχει ξεκινήσει με έναν έντονο ρυθμό τις επαφές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, μπορεί να μην ήταν όλοι παρόντες, αλλά ελπίζω ότι στην προηγούμενη συνάντησή μας, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα να, κάνουμε και άλλο, να οργανώσουμε και άλλη συνάντηση, και άλλο πάρτι. Λοιπόν, ευχαριστούμε και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε στις αρχές της Βελγικής, της Προεδρίας να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητές μας για την εσωτερική αγορά και για την προστασία των καταναλωτών. θα δείτε, ε, και το είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής, ότι στο πρόγραμμα εργασιών μας, το επόμενο εξάμεινο, έχουμε καθορίσει κάποιες προτεραιότητες, κάποιους στόχους που αφορούν την εσωτερική αγορά και την προστασία των καταναλωτών. Στην ομιλία μου θα επανέλθω σε κάποια σημεία, έξι θέματα πιο συγκεκριμένα, τα τρία που είναι ύψιστη της σημασίας για μένα. Το ένα είναι η βάνθηση τη απλώς της τη ε, αγοράς, της εσωτερικής αγοράς. Το δεύτερο αφορά την οδηγία για την προστασία των καταναλωτών. Και το τρίτο σημείο είναι η οδηγία για την καθυστέρηση των πληρωμών. Ε, ένα θέμα για το οποίο η Επιτροπή έχει αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο. Θα ξεκινήσω με το πιο σημαντικό στοιχείο, στα μάτια μου τουλάχιστον, που αφορά την περαιτέρω εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς. Πιστεύω ότι η χρηματοπιστωτική κρίση την οποία ζήσαμε πρόσφατα ε, έδειξε ότι το ευρωπαϊκό σύστημα υποφέρει από, κάποιες, από κάποια κενά. Και αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ευημερία μας και να έχουμε μια ανάπτυξη, θα πρέπει να γίνει μια σωστή ανακατανομή του πλούτου και να υιοθετήσουμε ένα μοντέλο το οποίο θα μας επιτρέψει να έχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει κάποιες προτεραιότητες, πρωτοβουλίες, έτσι ώστε αυτή η, ανάπτυξη να υπάρξει στην Ευρώπη ουσιαστικά πλέον. Και θα ήθελα να, κάνω μια ιστορική αναδρομή. Το 1992 όταν η Ευρώπη μετά από μια ανάπτυξη κάπως χαμηλή με την προεδρία του Ζακ Ντελόρ ξεκίνησε το μοντέλο αυτό, το μοντέλο αυτό της εσωτερικής αγοράς. Ε, τα πράγματα βελτιώθηκαν, ε, αποκτήσαμε πίστη και εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό μοντέλο, ε, το οποίο είναι πιο δυναμικό και νομίζω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε σε, αυτό το, σε αυτή την δυναμική του, της εποχής του Ζακ Ντελόρ. Μπορεί μεν οι περιστάσεις να είναι διαφορετικές, όμως η Ευρώπη είναι, έχει καθυστερήσει στα θέματα αυτά ε, σε σχέση με άλλες υπήρους και βλέπουμε ότι στην Ασία ή στην Νότιο Αμερική ε, έχουμε μια οικονομική ανάπτυξη, την οποία εμείς ε, ζηλεύουμε. Ο καθηγητής, ο κύριος Μάριο Μόντι, ο οποίος ήταν και πρώην επίτροπος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει, έκανε μια εξαιρετική δουλειά, δημοσίευσε ένα κείμενο, ε, στο οποίο ακριβώς διαπιστώνει την ε, κούραση που υπάρχει για αυτή την ολοκλήρωση, κούραση δηλαδή κόποση στην διαδικασία ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε κάποια συγκεκριμένα, κάποιες συγκεκριμένες προτεραιότητες και πρωτοβουλίες έτσι ώστε να καλυφθούν τα κενά. Και κάνει κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις για να βγούμε από το αδιέξοδο. Πιστεύω ότι σήμερα, χάρη στο νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο βιώνουμε στην Ευρώπη, δηλαδή χάρη στην συνθήκη της Λισαβόνας και χάρη στις αυξημένες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουμε την δυνατότητα, έχουμε την ευκαιρία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ακολουθήσει την Βελγική Προεδρία έτσι ώστε ε, να υλοποιηθεί ε, το κείμενο αυτό του Μάριο Μόντι, έτσι ώστε να έχουμε ένα πραγματικά νέο καινοτόμο πρόγραμμα. Ο Επίτροπος κ. Μπαγνιέ θέλει και αυτός ε, να ε, ε, καταλήξουμε σε μια single act ε, Single Market Act, σε μια πράξη ε, ενιαίας αγοράς. Αυτή την ε, πρόθεση την είδαμε και σε μια έκθεση Λεκλάρκη η οποία συζητήθηκε και υιοθετήθηκε και στην Επιτροπή σας. Αυτή η Single Market Act είναι μια φιλόδοξη πρόταση και ελπίζουμε ότι οι βιομηχανίες, οι οικονομικοί κύκλοι θα καταλάβουν την το, το διακύβευμα και θα κάνουν ό,τι μπορούν έτσι ώστε να υλοποιηθεί ουσιαστικά η ενιαία αγορά. Ε, ο Επίτροπος Μπαγνιέ ε, θέλει τον, στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου να συζητηθούν οι 30 προτάσεις που υποβάλλει η Κομισιό έτσι ώστε το 2012 να είμαστε έτοιμοι για να υλοποιήσουμε την ενιαία αγορά. 20 χρόνια δηλαδή ακριβώς μετά τα πρώτα βήματα του Ζακ Delors. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή προσοχή και στα θέματα καινοτομία και στη σημασία που έχει καινοτομία, διότι πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Καταρχά, στον τομέα της τυποποίηση. Ξέρω ότι ο πρόεδρο σα ε, ε, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα με την τυποποίηση, γιατί η τεχνολογική ανάπτυξη είναι τόσο γρήγορη τις, μέρε μα, ε, έτσι ώστε τα, οι στόχοι που θέτουμε εμεί στην Ευρώπη όσον αφορά την τυποποίηση κινδυνεύουν να, μείνουν, να είναι καθυστερημένη. Ε, δηλαδή η όλη Ευρώπη καθυστερεί σε σχέση με τους εταίρους της. Επίσης η σημασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Την προηγούμενη εβδομάδα η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων συζήτησε τα θέματα αυτά μαζί μου και τα, εγώ τους τόνισα την σημασία του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας διότι με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσουμε τις μεγάλες ε, εταιρείες, τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επίσης να ε, εποφεληθούν από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Και ξέρω ότι και η Επιτροπή σας ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για αυτά. Τρίτο σημείο, θα πρέπει να έχουμε ε, δημόσιες αγορές ε, οι οποίες να ενδιαφέρονται για τις καινοτομίες. Θα πρέπει να υιοθετήσουμε ένα πρόγραμμα εργασίας ε, όπου θα ασχολούμε όχι μόνο με την τιμή της εσωτερικής αγοράς αλλά και με την ποιότητά της. Αυτή η καινοτομία, η θα πρέπει να αποτελεί ένα σημαντικό, μια σημαντική πτυχή μιας οποιοδήποτε εσωτερικής αγοράς. Στις στις Βρυξέλλες θα, υιοθετήσουμε ένα, θα ε, οργανώσουμε ένα συνέδριο που αναφέρεται, που θα έχει σαν τίτλο From, From Knowledge to Competitiveness, από την γνώση στην ε, ανταγωνιστικότητα ε, και εκεί θα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Τα θέματα της ε, καινοτομία για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά, τα θέματα της καινοτομία και της ανταγωνιστικότητας. Βέβαια καταλαβαίνω ότι ανάλογα με την πολιτική οικογένεια που ανοίγει ο καθένας μπορεί από χρόνο να είναι διαφορετικές, όμως μια σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς είναι ζωτική σημασία για όλους μας και χρειάζεται μια καινούργια ανάγκη αυτή, αυτή η αγορά. Πρέπει κάτι να κάνουμε, κάτι καινοτόμο. Επίσης, άλλο σημείο, η οδηγία για το δίκαιο των καταναλωτών. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί συνάντησα κάποιου βουλευτέ που έχουν που έχουν αφιερώσει αρκετό χρόνο, Ο κύριο Βάμπ, επίση υπάρχουν και σκιώδει συζητητέ που ασχολούνται με όλα αυτά τα θέματα και ξέρω ότι και η Επιτροπή σα έχει αφιερώσει πάρα πολλέ ε, συνεδριάσει ε, για τα θέματα αυτά του δικαίου των καταναλωτών. Ε, επίση στο Συμβούλιο 43 συνεδριάσεις έχουν αφιερωθεί για αυτό το θέμα. Γιατί είναι σημαντικό τώρα αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό διότι πιστεύω ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών αποτελούν τον πυρήνα της εσωτερική αγοράς. Εάν θέλουμε πραγματικά οι καταναλωτές να έχουν εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις ε, της Ευρώπης, θα πρέπει η οδηγία αυτή για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών να είναι μια ισορροπημένη οδηγία. Και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε ο φάκελος αυτό να προχωρήσει. Ε, θα ακούσατε επίσης ε, ότι η Επίτροπος, η κυρία Βίβιαν Ρέ, Ρέντινγκ υπογράμμισε την ε, σημασία του θέματος αυτού και ε, επίσης ε, μίλησε και για την στοχευμένη μέγιστη εναρμόνιση που θα πρέπει να υιοθετηθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα... να λάβουμε υπόψη μας ότι για ιστορικούς λόγους τα 27 κράτη-μέλη έχουν διαφορετική όραμα, διαφορετική προοπτική, διότι και διαφορετική εξέλιξή τους. Όμως εμείς σαν Προεδρία θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, πλαισιώσουμε και να αντιμετωπίσουμε το, το πρόβλημα με έναν ε, αντικειμενικό τρόπο. Θα πρέπει για κάθε κεφάλαιο να δούμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία και για την αγορά και για τους καταναλωτές και να πετύχουν σε τον περισσότερη εναρμόνιση. Ο στόχος μας μπορεί να είναι φιλόδοξος μεν, αλλά ελπίζουμε ότι μέχρι το, την σύνοδο κορυφής ε, του Δεκεμβρίου, του 2010, δηλαδή να έχουμε κάποιες συγκεκριμένες ε, ε, προτάσεις για την οδηγία. Και ελπίζουμε, Πρόεδρε, ε, και η δική σας Επιτροπή να πει την άποψή της για τον φάκελο αυτό, έτσι ώστε στην επόμενη Προεδρία, την Ουγγρική Προεδρία, να επικυρώσουμε την, να υιοθετήσουμε την οδηγία επίσημα. Όμως, πέραν της οδηγίας για την προστασία των καταναλωτών, θα πρέπει να έχουμε και μια ουσιαστική προστασία του καταναλωτή και κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας 22 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες σε συνεργασία με τον Επίτροπο Τζον Ντάλι θα οργανώσουμε μια ημερίδα για την προστασία του Ευρωπαίου καταναλωτή, έτσι ώστε να υπογραμμίσουμε τη συνεργασία ανάμεσα στις 27 ε, υπηρεσίες ελέγχου ε, και παρακολούθησης, έτσι ώστε να έχουμε έναν μια σωστή εναρμόνιση ε, και μια σωστή λειτουργία των όλων υπηρεσιών ε, παρακολούθησης και επίβλεψης. Εμείς στο Βέλγιο έχουμε μια υπηρεσία αντίστοιχη και ξέρουμε ακριβώς επειδή ε, παρακολουθούμε το θέμα ότι υπάρχουν προβλήματα και στη συνεργασία ανάμεσα στις χώρες και αυτά τα προβλήματα πρέπει να τα λύσουμε. Γι' αυτό θα πρέπει οι υπηρεσίες των 27 ε, κρατών μελών να μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά και τις επιχειρήσεις και, τις, ε, και τους καταναλωτές. Ένα άλλο θέμα πάρα πολύ σημαντικό είναι η οδηγία για την καθυστέρηση των πληρωμών. Ξέρετε ότι η χρηματοπιστωτική ε, κρίση την οποία ζούμε έφερε σε δύσκολη θέση κάποιες επιχειρήσεις. Ε, σύμφωνα με τον δίκτυο Ευρωπαίων ε, Πληρωμών για το 2006, η καθυστέρηση είναι στην Ευρώπη είναι 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα τεράστιο ποσό δηλαδή και αυτό το ποσό αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην, ε, στην Ευρώπη. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση και η Επιτροπή ΙΜΚΟ και η κυρία Βάιλερ, η συγγήτρια, πραγματικά έκαναν εξαιρετική δουλειά στην, ε, δηλαδή στην προσπά, στις σας για να καταλήξουμε σε ένα πλαίσιο συμφωνίας ανάμεσα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τις ε, ε διοικητικές υπηρεσίες έτσι ώστε να έχουμε κάποια, κάποιες ε, διατάξεις, κάποιες κοινέ προθεσμίες έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μην αποτελούν τα θύματα αυτής της, αυτών των καθυστερημένων πληρωμών. Τώρα, μια και γνωρίζουμε και τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ελπίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της Βελικής Προεδρίας θα, αναλάβουμε, θα, θα μας αναθέσει μάλλον το Συμβούλιο μία εντολή ε, να ξεκινήσει ένας τρίλογος κατά τη διάρκεια της Βελικής Προεδρίας έτσι ώστε να ξεκινήσει μία ανάγνωση του σχεδίου αυτού ε, παρουσία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, κάποια σημεία έντασης, ε, κυρίως αναφορά την ε, διαφορά ανάμεσα, αντιμετώπιση ανάμεσα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τις δημόσιες επιχειρήσεις, ε, ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε την μέγιστη προθεσμία των 60 ημερών, οι ιατρικές υπηρεσίες που θα πρέπει και αυτές να αποτελέσουν ένα κομμάτι. Τέλος πάντων, παρά αυτά τα εμπόδια, πιστεύω ότι από την αρχή της προεδρίες μας έχουμε κάνει καλή δουλειά και στο Συμβούλιο υπάρχει ένα σχέδιο συμφωνίας, έχει, διαγράφεται ένα σχέδιο συμφωνίας και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε κάποια οριστική λύση τον, το φθινόπωρο. Το Κοινοβούλιο επίσης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά πάνω στο θέμα και από εδώ και πέρα τώρα θα πρέπει το Συμβούλιο να αναλάβει την δέσμευση, να υλοποιήσει όλες αυτές τις υποσχέσεις θα ήθελα να θίξω επίσης ε, και κάποια άλλα θέματα τα οποία για μα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Παραδείγματο χάρη το θέμα της εναρμόνισης των οικοδομικών υλικών και των κλωστοφαντουργικών ε, Έχουμε, ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί και εσείς με αυτό το θέμα και θέλουμε να ε, επιταχυνθεί η διαδικασία της ανάγνωσης του κειμένου κατά διάρκεια της ε, Προεδρίας μας. Ξέρουμε ότι η κλωστοϊφαντουργία και ο κατασκευαστικός τομέας είναι ε, ζωτική σημασία για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς. Είναι πάρα πολύ σημαντική τομή για όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτά τα θέματα πρέπει να προχωρήσουμε. Επίση, τα τυχερά παιχνίδια. Ένα άλλο θέμα που μα απασχολεί. Η Βελγική Προεδρία είναι ιδιαίτερα χαρούμενη διότι έχει, έχει δημοσιεύσει η Επιτροπή, η Κομισιό, αυτό, αυτή την πράσινη βίβλο για τα τυχερά παιχνίδια και θα γίνει και μια συζήτηση επίσης στο Συμβούλιο για τα online τυχερά παιχνίδια ε, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Επίσης, ένα άλλο θέμα αφορά το λιανεμπόριο. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για πολλά κράτη-μέλη πριν από 15 μέρες περίπου υιοθετήσαμε ένα κείμενο για τα δυνατά σημεία και για τις αδυναμίες του λιανεμπορίου και θα ήθελα να ασχοληθώ τώρα αυτή τη στιγμή με τις αδυναμίες του λιανεμπορίου διότι η πολιτική τις αδυναμίες πρέπει να υπογραμμίζουν και να προσπαθούν να βρουν μια λύση. Ε, βέβαια η παραγωγικότητα είναι πολύ χαμηλότερη στην Ευρώπη σε σχέση με τις ΗΠΑ. Μια άλλη ε, αδυναμία είναι μια έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τις τιμές για κάποια προϊόντα όπου, εκεί, όπου τα περιθώρια κέρδους είναι τεράστια στο λιανεμπόριο. Επίσης είναι ένα θέμα της κυριαρχίας της αγοράς από κάποιους φορείς, από κάποιες αλυσίδες διανομής προϊόντων ε, και πολλές φορές αυτά τα περιθώρια κέρδους είναι τεράστια και δεν υπάρχει διαφάνεια ταυτόχρονα. Επίσης, ε, τα, ε, τα πρότυπα είναι τόσο υψηλά που οι νέοι, οι καινούργοι στην αγορά δεν μπορούν να βρουν τη θέση τους και δεν θα πρέπει οι καταναλωτές να αποτελούν θύματα των υψηλών τιμών που εφαρμόζουν κάποιοι κλάδοι. Η μελέτη αυτή της ε, Κομισιόν είναι πολύ ενδιαφέρουσα, θα την μελετήσουμε, θα τη συζητήσουμε και στο Συμβούλιο της Ανταγωνιστικότητα του Δεκεμβρίου 2010 και ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, πριν ολοκληρώσω θα ήθελα να σας πω δύο πράγματα. Καταρχάς ξέρω ότι θα υπάρχει μια πρώτη έκδοση πιλότος και χάρη στην ε, Επιτροπή ΙΜΚΟ για την ε, εσωτερική αγορά της τη συνάντηση της 9ης Νοεμβρίου για την εσωτερική αγορά. Και ξέρω ότι πάρα πολλά μέλη της Επιτροπής σας θεωρούν ότι αυτή η συνάντηση είναι πάρα πολύ σημαντική και θα ήθελα να σας ε, υποσχεθώ ότι θα σας υποστηρίξουμε για αυτό το φόρουμ με όλες μας τις δυνάμεις. Επίσης θα ήθελα να σας προσκαλέσω σε μια επίσκεψη εργασίας στο Βέλγιο. Ακόμα δεν έχουμε ορίσει ημερομηνίε, αλλά περιμένουμε την ε, Επιτροπή ΙΜΚΟ έτσι ώστε να μπορούμε να επισκεφθούμε επιτόπου τα σημεία και να συζητήσουμε ποια είναι τα σημεία ε, που αφορούν την καλύτερη λειτουργία της ουσιαστικής αγοράς. Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο το οποίο έχουμε ξεκινήσει ε, και θέλουμε επίσης να εξασφαλίσουμε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, Ξέρω ότι και η δική σας Επιτροπή είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη και θέλει να βελτιώσει γενικά το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και σε μένα να βλέπετε έναν σύμμαχο στις προσπάθειές σας. Διότι και εγώ θα ήθελα ε, αυτός ο νέος ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενισχυθεί, διότι εμείς σεβόμαστε τις αυξημένες αρμοδιότητες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ελπίζουμε ότι τους επόμενους έξι μήνες ε, θα έχω την ευκαιρία να σας ξανασυναντήσω, ε, να τα πούμε, να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε ε, κάποια θέματα και κάποιους φακέλους και να καταλήξουμε σε, κάποια συμφωνία. Αυτά κύριε Πρόεδρε, είμαι στη διάθεσή σας ε, για να απαντήσω στις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής. Ερωτήσεις ε, που αφορούν που, όχι μονάχα τα θέματα τα οποία έθιξα, αλλά ό,τι άλλο πρόβλημα, θέμα θέλετε να θίξετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Uh, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ για την πλήρη παρουσίαση και επισκόπηση που μας δώσατε και είναι σαφές ότι έχετε ήδη βαθιά γνώση των θεμάτων και βαθιές πεπιθήσεις σε σχέση με τη σημασία των εκθέσεών μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το χαιρετίζει η Επιτροπή μας γιατί είμαστε πάρα πολύ φιλόδοξοι, θέλουμε πράγματι να προχωρήσουμε στα θέματα αυτά. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το οποίο είπατε και η σημασία που δώσατε στα θέματα της, του λιανεμπορίου γιατί εμείς έχουμε ήδη αποφασίσει στην Επιτροπή μας να κάνουμε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας σε σχέση, σε απάντηση μάλλον, του εγγράφου της ε, Κομισιόν. Στις 10 Δεκεμβρίου πιστεύω ότι αυτό το θέμα θα μπορέσει να εγερθεί στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και ελπίζουμε ότι θα έχουμε τελειώσει αυτή την έκθεση. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να δώσουμε και εμείς τη δική μας συνεισφορά και ίσως και ο εισηγητής μας θα μπορέσει να σας δώσει τα πορίσματα αυτής της έκθεσης. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι χρήσιμο. Επίσης ήμουν παρόν στο πρόσφατο Συμβουλίο Ανταγωνιστικότητας που ήσασταν και εσείς παρόν για να παρουσιάσω την έκθεσή μας για την ενιαία αγορά, την έκθεση του κυρίου Γκρέκ. Πιστεύουμε, κρέσου, πιστεύουμε, δεν νομίζω ότι ήταν στο αρχικό σας πρόγραμμα, αλλά πιστεύω ότι ο κύριος Μπαρνιέ θέλει τον Οκτώβριο να παρουσιάσει και αυτό τις ιδέες του για ένα νομοθέτημα για την ενιαία αγορά, που είναι φυσικά μια ευκαιρία και για σας να συμβάλλεται στην διαμόρφωση αυτού του νομικού πλαισίου. Στις 9 Νοεμβρίου θα έχουμε αυτή την εκδήλωση η οποία θα είναι πολύ σημαντική για την πρόθεση και τις διαδικασίες της νομοθετικής για την ε, νομοθετική πράξη για την ενιαία αγορά. Αυτό πιστεύω λοιπόν θα μπορέσει να δημιουργήσει ένα μεγάλο αντίκτυπο αν υπάρξει η συνεργασία και των τριών κυρίων θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά υπομορφή λοιπόν εισαγωγή από μένα. Τώρα περνάω στου συναδέλφου. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στου εκπροσώπου τεσσάρων πολιτικών κομμάτων και μετά μπορείτε να απαντήσετε. Αυτός είναι ο πρώτο γύρος, Σουάμπ, Ταραμπέλα, Ροσφόρ, και ο κύριος Τρενταφυλλίδης και θα ακολουθήσει ένας γύρος με την κυρία Βανιό, τον κύριο Κουρέα Δικάμπους και την κυρία Βάιλα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θέλει να λάβει το λόγο. Μπορεί να επανέλθει σε ένα μεταγενέστερο γύρο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον κύριο Σουάμπ. Σας ευχαριστώ. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε ε, Υπουργέ, εμφανιστήκατε στο Στρασβούργο. Από την Ισπανική Προεδρία έχει περισσέψει αρκετή δουλειά. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι η Βελική Προεδρία μπορεί να γίνει μια επιτυχία. Όπως είπατε και όπως φέρατε και το παράδειγμα του Ζακτελόρ στη δεκαετία του 90 που επανέφερε ένα δυναμισμό Φαίνεται πάντω στο Συμβούλιο μην υπάρχει πάντοτε αυτό το πνεύμα. Εάν μπορεί η Βελγική Προεδρία να το προωθήσει τόσο το καλύτερο. Αναφέρατε ορισμένα θέματα στα οποία θα κάνετε μια προσπάθεια. Αυτό βεβαίω θα είναι επωφελέ για όλου μα, και για εσά και για εμά και για του καταναλωτέ. Αναφερθήκατε σε ορισμένε οδηγίε. Θα θίξω κυρίω τι δύο που εκκρεμούν και ενώπιον του Συμβουλίου για τι καθυστερήσει πληρωμών αφενός με αρκετά διακομματικό τρόπο διείδαμε τον κίνδυνο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα αναπτυχθεί ένας ανταγωνισμό για το ποιοι τομεί θα εξαιρεθούν από την οδηγία καθυστέρηση πληρωμών. Χρειαζόμαστε όμω ένα ανώτατο όριο για τις συμβάσεις B2B. Η ερώτησή μου είναι, θεωρείτε ότι η διαπραγματευτική εντολή που ενέκρινε το Συμβούλιο και πιστεύω θα το θα το, θέσει το θέμα αυτό και η κυρία Βάιλερ μετά. Μπορούμε να αναμένουμε λοιπόν ότι θα υπάρξει πρόοδο στο θέμα. Ή είναι περισσότερο μια προσπάθεια να καλυφθούν οι διαφορές απόψεων. Δεύτερον, η οδηγία για την προστασία των καταναλωτών. Είπατε με αρκετά φιλόδοξο τρόπο ότι μέχρι τέλους του έτους θα υποβάλλεται ολοκληρωμένη πρόταση Έχω γράψει μάλιστα τη λέξη ολοκληρωμένη εδώ στι σημειώσει μου. Την προηγούμενη εβδομάδα με τους κοιότητε συγητέ, συναντηθήκαμε με του πρόεδρου των Επιτροπών για να συζητήσουμε την στρατηγική μα την στρατηγική μας προσέγγιση. Σημειώθηκαν ορισμένε αποκλήσεις απόψεων. Θα είδατε κι εσείς ήδη ότι η δική μου άποψη είναι κυρίως ότι μέσα στα πλαίσια αυτής της θεώρησης από τη σκοπιά της ε, ενίας αγοράς θα πρέπει να προωθήσουμε μια κοινότητα στόχων αλλά στους τομείς εκείνους όπου είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Η Βελγική Προεδρία με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίσει το θέμα της ενοποίησης στην οδηγία. Το έχετε ήδη συζητήσει αυτό στο Συμβούλιο. Μπορείτε να πείτε λίγα λόγια για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να είναι ο βασικός στόχος μια ενοποίηση ή να αρκεστείτε περισσότερο στην απολύτως απαραίτητη εναρμόνιση. Ευχαριστώ κύριε Σφάβο. Κύριο Ταραμπέλα. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ στην Επιτροπή μας. Και τώρα φυσικά θα γυρίσω στα γαλλικά, όπως φαντάζεστε. Έχετε αναφερθεί σε ορισμένα θέματα, σε ορισμένους φακέλους που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε μαζί αλλά βλέπω ότι στο πρόγραμμα της Βελικής Προεδρίας για την συμπλήρωση της ε, εσωτερικής αγοράς βλέπω να υπάρχει λίγη κινητικότητα σε συγκεκριμένους τομείς που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τους πολίτες μας και θα ήθελα η Βελική Προεδρία να ασχοληθεί περισσότερο με την πρωτοβουλία της Κομισιόν σε σχέση με τις υπηρεσίες κοινοφελούς χαρακτήρα. Μήπως θα θεωρούσατε λοιπόν κύριε Υπουργέ ότι η Προεδρία θα μπορούσε να είναι πιο φιλελεύθερη όπως και στην περίπτωση της αγοράς ηλεκτρισμού και στην αγορά τηλεπικοινωνίας. Διότι στις περιπτώσεις αυτές εκεί δεν υπήρξε πραγματική μείωση για τον καταναλωτή παρά την σπουδή της Κομισιόν. Ακόμα και η ποιότητα των υπηρεσιών δεν μπορούμε να πούμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις αυτές βελτιώθηκε. Μήπω πιστεύετε λοιπόν κύριε Υπουργέ ότι αντί να προχωρείτε σε τέτοιες βεβαιασμένε ενέργειες, αντί να κάνετε κάτι τέτοιο, μήπως θα έπρεπε να αναλύσετε με πιο ενεργητικό τρόπο τα αποτελέσματα, τα αντικειμενικά αποτελέσματα, ίσως θετικά αποτελέσματα εν μέρη, αλλά και τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν στη φιλελευθερωποίηση στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό, την επιλογή, τη δυνατότητα επιλογής, την ποιότητα και τις τιμέ για του καταναλωτές. Η δική μα ομάδα έχει ζητήσει επανειλημμένα να υπάρχει ένα χάρτης ενέργειας για τους καταναλωτές με την πρωτοβουλία και τη κυρία Βίτς στο παρελθόν και είχε υποσχεθεί η Κομισιόν ότι θα υπάρξει μια τέτοια χάρτα αλλά αυτό δεν έγινε δεκτό διότι το απέρριψε το Συμβούλιο κατ' πίεση του Κοινοβουλίου και εσείς αναφερθήκατε στο ρόλο του Κοινοβουλίου, καταφέραμε εμείς να έχουμε μια μείωση του, των τιμών περιαγωγής στην κινητή τηλεφωνία. Αυτό ήταν μια απόφαση η οποία επετεύχθη χάρη στην επιμονή του Κοινοβουλίου και επίσης τη χρήση του διαδικτύου σε περιαγωγή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως θα μπορούσε το Συμβούλιο να πιέσει την Κομισιόν για να υπάρξει και μια ενοποίηση των τιμών που είναι ακόμα πάρα πολύ μεγάλη ψαλίδα τους, ένα προς οκτώ κάτι το οποίο δεν δικαιολογείται από τον ανταγωνισμό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Τάραμπελ. Ο κύριος Ροσφόρ. Σας ευχαριστώ. Θέλω να σας συγχαρώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ μάλλον, γιατί τα λόγια σας καταδεικνύουν ότι έχετε ήδη εισέλθει πλήρως στα θέματα αυτά. Έχετε αναφέρει ποια είναι τα κύρια θέματα που σας απασχολούν, τα οποία επικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό με τις δικές μας ανησυχίες και τα ενδιαφέροντά μας. Συμφωνούμε ίσως όλοι μας για τις γενικές κατευθυντήρες γραμμές που θέλουμε να θέσουμε στα διάφορα κεφάλαια. Φυσικά στη συνέχεια είναι το πρακτέο, πώς θα μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά. Έχετε δίκιο επίσης να ακολουθείτε μια συγκεκριμένη σειρά στον τρόπο προσέγγισης για τα θέματα αυτά. Πιστεύω παραδείγματος χάρη ότι όταν αναφέρεστε στην ανάκαμψη της εσωτερικής αγοράς και εγώ αντίθετα τον κύριο Ταραμπέλα μιλάω για ανάκαμψη και όχι για συμπλήρωση, για ε, ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, νομίζω ποτέ δεν θα είναι απόλυτα ολοκληρωμένη αυτή η αγορά, ήταν πολύ σωστό αυτό που αναφερθήκατε στη σημαντική έκθεση του κυρίου Μόντι. Νομίζω ότι όλοι αλλάζουν, ο Μάριο Μόντι που είχα γνωρίσει πριν από 4-5 χρόνια είναι διαφορετικός από το σημερινό Μάριο Μόντι. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος όπως ο κύριος Μόντι αλλάζει την άποψή του με αυτόν τον τρόπο και εξελίσσεται και πρόκειται για ένα άτομο με πολύ βαθιά εδρεωμένη εμπειρία, νομίζω ότι μπορούμε να κατανοήσουμε ότι το New Deal, η νέα οργάνωση των πραγμάτων που προτείνει, είναι αποκύημα διαπραγματεύσεων και συνεννοήσεων με τα κράτη-μέλη. Και μιλώ για τα κράτη-μέλη γιατί μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πω προς το Συμβούλιο ότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία αντιδρούν και χρονοτριβούν για να εφαρμοστούν οι προτάσεις του Μάριο Μόντι. Το μπαλάκι βρίσκεται πράγματι στο, γήπεδο, στο τμήμα του γήπεδου του Συμβουλίου και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια σειρά προτάσεων για τη βελτίωση τη εσωτερική αγορά και είμαι σίγουρο ότι ο κύριο Μπαρνιέ από την Κομισιόν θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό, αλλά το πνεύμα τη έκθεση Μόντι πιστεύω ότι είναι πιο ισχυρό από τι προτάσει που μπορούν να προέλθουν μεμονωμένα και εφόσον υπάρχει αυτή η πρόβλεψη για ένα νομοθετικό κείμενο, αυτή η πράξη για την ενιαία αγορά, αυτό το νομοθέτημα για την ενιαία αγορά θα είναι πραγματικά κάτι το οποίο θα προωθήσει το κοινοτικό πνεύμα ένα βήμα πιο πέρα ή θα είναι μια σειρά από περιορισμένες εμβέλειες διατάξεις. Ένα δεύτερο στοιχείο, εσείς αναφερθήκατε κύριε Υπουργέ, στην οδηγία για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Συμφωνούμε όλοι εδώ και ελπίζω ότι θα μπορέσω να συνεδριθώ και με τον εισηγητή τον κύριο Σουάμπ. Ελπίζουμε ότι η Βελική Προεδρία θα μπορέσει να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα και να φτάσουμε σε μια πρώτη συμφωνία. Αλλά θα ήθελα πω σχετικά ότι η διατύπωση η οποία υπάρχει μέσα στο πρόγραμμα της Βελικής Προεδρίας μου φαίνεται ότι είναι μια κάπως υπαναχώρηση σε, αυτά, σε σχέση με αυτά που είχαν προταθεί στο παρελθόν, ακόμα και σε σχέση με αυτά τα οποία είπατε εσείς. Είναι μια ασαφής διατύπωση. Λέτε ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε υψηλή προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Αυτό είναι σχεδόν μια αμυντική στάση. Λες και απλώς πρέπει να φροντίσουμε να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας που ήδη υπάρχει. Αν θέλετε να κινητοποιήσετε τους καταναλωτές θα πρέπει να πείτε κάτι περισσότερο, να υπάρχει μια εγγύηση του τωρινού επίπεδου προστασίας των καταναλωτών και για μια σειρά νέα θέματα θα υπάρξει και βελτίωση των δικαιωμάτων τους, λαμβάνοντας υπόψη τους νέους κανόνες της αγοράς και ιδίως το ηλεκτρονικό εμπόριο. Είπατε ότι ήσασταν παρόν σε 43 συνεδριάσεις για τα θέματα αυτά. Εμείς έχουμε καθυστερήσει, αλλά θα σας προλάβουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Και τέλος, νομίζω ότι έχετε δίκιο να μιλάτε για θέματα όπως η καθυστέρηση πληρωμών. Η ομάδα μου υπογραμμίζει τη σημασία αυτού του θέματος, όπως και του Ευρωπαϊκού Διπλώματος ε, Τεχνίας, που είναι κεφαλαίωρες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αναφερθήκαμε στο θέμα αυτό πολλές φορές και ζητούμε αδειμόνως να προχωρήσει πιο πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έρχομαι και πάλι στο ερώτημα του κυρίου Σουάμπ. Η πλήρης στοχευμένη εναρμόνιση που αναφέρατε προηγουμένως, αναφερόμενος στα λόγια του κυρίου Επιτρόπου, ποια είναι η θέση του Συμβουλίου. Θα πρέπει να είναι εξελαχίστων αυτή η εναρμόνιση και υπάρχει μια δυνατότητα μικτής εναρμόνισης η οποία δεν θα είναι ούτε πλήρης ούτε μια εκ των ελαχίστων εναρμόνιση. Κάτι το οποίο θα μείωνε σημαντικά τις φιλοδοξίες μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φιλιππίδη, Φιλίδης. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε και εσείς αλλά και προλαλήσαντε συνάδελφοι στην έκθεση Μόντι μια ε, πολύ εμπεριστατωμένη μελέτη θα έλεγα και ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσον ασπάζεστε αυτά τα οποία προτείνει ή κατά πόσον έχετε δημιουργήσει κάποια εντύπωση για πιθανές αλλαγές που μπορείτε να εισηγηθείτε και ποιες θα είναι αυτές οι αλλαγές. Επίσης, ο κύριος Μόντι σε προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής μας εδώ, ε, αναλύοντας τις ενέργειες που πρέπει να αναλυφθούν για την υλοποίηση της έκθεσης του για την νέα, νέα ενιαία αγορά, κάλεσε τον πρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Μπαρόσο, να αναλάβει προσωπικά το θέμα, ώστε ο συντονισμός εντός της Κομισιόν να προέλθει από το ανώτατο επίπεδο. Εσείς ως Προεδρία τώρα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αναλαμβάνετε πρώτοι αυτό το εχείρημα της υλοποίησης των συστάσεων Μόντι. Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα αναλάβετε εντός του Συμβουλίου. Έχετε κάποιες ενέργειες που μπορείτε να μας συζητηθείτε. Ευχαριστώ. Thank you very much. Um, I'll ask the Minister then to respond to, uh, to the first four points and then we'll take... Uh, θα δώσω το λόγο τώρα στον Υπουργό να απαντήσει στα τέσσερα πρώτα, τέσσερις πρώτες ερωτήσεις και μετά θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος ερωτήσεων. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και για τα εισαγωγικά λόγια που είπατε. Ε, για τα όσα είπατε για τις εκθέσεις που ήδη διεκπεραιώνονται στην Επιτροπή σας και για τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεστε να συνεργαστείτε με το Συμβούλιο. Για τον τομέα του λιανικού εμπορίου νομίζω θα μπορέσουμε μέχρι το Δεκέμβριο να συντάξουμε συμπεράσματα και θα μας διευκολύνει εάν μπορέσει να συμβαδίσει η προσπάθεια αυτή με την έκθεση της Επιτροπής σας. Χρειάζεται λοιπόν να εναρμονίσουμε τα χρονοδιαγράμματά μας και ελπίζω ότι αυτό είναι δυνατόν. Απαντώ στον κύριο Σφάμπ που με ρώτησε για τις καθυστερήσεις πληρωμών και πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα. Είναι όντως η πρόθεσή μας στο Συμβούλιο να ζητήσουμε και να λάβουμε διαπραγματευτική εντολή για την διεξαγωγή τριμερούς διαλόγου με το Συμβούλιο ω φελική Προεδρία, ώστε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό σχετικά με το ποιοι τομεί θα καλύπτονται από την οδηγία. Και εμά μας ενδιαφέρει το B2B, το business to business που είπατε πριν, γιατί έχουμε την φιλοδοξία να προστατεύσουμε και τις μικρές επιχειρήσεις. Μέσα λοιπόν στο Συμβούλιο αναζητούμε μια πλατφόρμα για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τη συζήτηση με το Κοινοβούλιο ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία μέχρι τέλους του έτους. Ο κ. Φάμπ με ρώτησε επίσης σχετικά με την εναρμόνιση. Με ρώτησε δηλαδή σχετικά με, την με το τελευταίο συμβούλιο υπό Ισπανική Προεδρία, όπου διαπίστωσε ότι μια μεγάλη πλειοψηφία των χωρών μελών τίνει προς μια μέγιστη εναρμόνιση, στοχευμένη. Αυτός είναι ο στόχος μας εν τέλει. Αλλά η προσέγγιση αυτή πρέπει να είναι ρεαλιστική. Ανάγνωση κεφαλαίου ανακεφάλαιο, ώστε να δούμε σε ποιες συμβαστικές λύσεις μπορούμε να καταλήξουμε, ώστε εν τέλει, στο τέλος της συζητήσεως δηλαδή, να δούμε πού μπορούμε να καταλήξουμε. Γιατί και το συμφέρον του του είναι σημαντικό, το ανέφερε ο κ. Ροσφόρ, αλλά βέβαια πρέπει να παραμείνουμε στο δυνατόν πιο εύκαμπτοι, πιο ευέλικτοι και στην διεξαγωγή διαμεθοριακών συναλλαγών, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη στην Ευρώπη. Με ρωτήσατε επίσης κύριε Σφάπ, μάλλον ε, ε, διάβασα προσεκτικά τα όσα είπατε για το άρθρο 4 της οδηγίας, όπου τονίσατε ότι η εναρμόνιση πρέπει να είναι στοχευμένη. Δεν θέλω να προκαταλάβω την συζήτηση που θα διεξαρθεί στο ε, Συμβούλιο. Νομίζω ότι παρά τις 3.43 λοιπόν αυτές ε, συνεδριάσεις είναι ενδιαφέροντα αυτά τα οποία αναφέρατε εσείς και μπορούμε να τα συζητήσουμε και περαιτέρω στο Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις υπηρεσίες γενικού, κοινοφελούς μάλλον χαρακτήρα, Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση η οποία μπορεί να έχει και ιδεολογική χρειά και είναι σημαντικό βέβαια να κάνουμε αυτή τη συζήτηση γιατί η πολιτική εμπεριέχει την ιδεολογία και είναι πολλές φορές αντιπαράθεση διαφορετικών ιδεολογικών θέσεων και χαίρομαι πάρα πολύ που θέσατε αυτό το θέμα. Εγώ υπάρχει φυσικά η βάση του άρθρου 14 στη συνθήκη της Λισαβόνας και το πρωτόκολλο 26. Εγώ διάβασα πολύ προσεκτικά την έκθεση του Μάριο Μόντι είδα σε ορισμένου τομεί, σε πολύ συγκεκριμένου τομεί, ιδίω σε ό,τι αφορά τα θέματα των τηλεπικοινωνιών, στον τομέα των τραπεζικών υπηρεσιών, στον τομέα των μεταφορών επίση. Αναφέρεται ο κύριο Μόντι στι απαραίτητε πρωτοβουλίε οι οποίε θα πρέπει να αναπτυχθούν για να ενισχυθούν αυτέ οι υπηρεσίε. Πιστεύω λοιπόν ότι ενώπιον τη συζήτηση που θα λάβει η χώρα στου κόλπου του Συμβουλίου ενώπιον και των πρωτοβουλίων του κυρίου Μπαρνιέ του αρμόδιου επιτό, αλλά φυσικά και λαμβάνοντα υπόψη την σημασία που αποδίδεται το θέμα αυτό, για μένα θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε σε ποιο συγκεκριμένο τομέα θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Παραδείγματο χάρη στο Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίε σε ό,τι αφορά τις ευρωζωνικές υπηρεσίε. Γιατί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μα να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ήπειρο στην οποία ένα τμήμα του πληθυσμού μονάχα έχει πρόσβαση σε ευρωζωνικές υπηρεσίες και άλλοι όχι. Αυτό είναι μια πολύ ευαίσθητη συζήτηση στα κράτη-μέλη μας. Νομίζω λοιπόν στο θέμα αυτό προφανώς θα αναμείνουμε τις ε, πρωτοβουλίες της Κομισιόν αλλά με μια στεναρή θέληση να προχωρήσουμε. <clears throat> Δεύτερον, θέσατε το ερώτημα για την περιαγωγή δεδομένων. Θα υπάρξει μια ενδιάμεση αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Προεδρίας μας. Δεν σας αποκρύπτω βέβαια ότι λόγω των πρωτοβουλίων που έχει αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που σας δίνει η Συνδίκη της Λισαβόνας θα πρέπει νωρίτερα και όχι αργότερα να, να αποφύγουμε τις εκπλήξεις των λεγόμενων λογαριασμών σφαλιάρα που μπορεί να φτάσει κάποιος σε, να πληρώσει ένα λογαριασμό 10.000 ευρώ χωρίς να το έχει αντιληφθεί. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για την Προεδρία μας να αναλάβει μια πρωτοβουλία και από τη δική σας πλευρά, την πλευρά του Κοινοβουλίου, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει αποφυγή αυτών των καταστάσεων. Κύριε Ροσουά, αναφερθήκατε στο New Deal του κυρίου Μόντι. Και όπως είπατε αυτό θα πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από μια απαρίθμηση πρωτοβουλειών όπως αυτές που ανέφερε και ο κύριος Μπαρνιέ. Η απόψη μου εδώ είναι πάρα πολύ σαφής. Πιστεύω ότι πρώτον θα πρέπει να προχωρήσουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο για τα θέματα αυτά, αλλά ακολουθώντας και κάποιο οδηγό πνεύμα. Δεν μπορούμε να έχουμε απλώς ένα κατάλογο σε τεχνικό επίπεδο. Θα πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο πνεύμα σε σχέση με την εσωτερική αγορά. Και διάβασα την έκθεση Γκρέκ, η οποία που αναφέρει τα προβλήματα των πολιτών όταν έχουν να κάνουν με διαμεθοριακές συναλλαγές. Και κατά την άποψή μου εδώ εμπλέκεται η ευθύνη και του Κοινοβουλίου <clears throat> αλλά και της Προεδρίας να βρίσκεται αυτό το σημείο πάντα σε προεξάρχουσα θέση και να προσπαθήσουμε να συγκεκριμενοποιήσουμε τις λύσεις παραμένοντας πάντα φιλόδοξοι. Γιατί η πεποίθησή μου είναι ότι αν η Ευρώπη θέλει να επιτύχει μεγαλύτερη ολοκλήρωση, αν η Ευρώπη θέλει να γίνει και πάλι ένα όραμα το οποίο υποστηρίζουν οι πολίτες της, είναι η ικανότητα ηγεσία των ανδρών και των γυναικών που βρίσκονται στο πολιτικό στερέωμα στην Ευρώπη. Από εκεί θα εξαρτηθεί λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία και αυτό το όραμα. Γι' αυτό θέλω να υπάρχει ένα άτομο το οποίο προσωποποιεί αυτήν την ε, πρωτοβουλία. Και δεν είναι τυχαίο που αναφέρουμε στον κύριο Ντελόρ. Όταν, υπήρχε, όταν έγινε η πρόταση για την έννοια αγορά ήμουν 19 χρονών. Έμπαινα μόλι στο πανεπιστήμιο. Και σας ε, διαβεβαιώ ότι τα χρόνια εκείνα η Ευρώπη φαινόταν να έχει ένα πνεύμα, μια φιλοδοξία αυτό είναι απαραίτητο να το έχει και πάλι σήμερα. Και εσείς μαζί με τους συναδέλφους σας θα πρέπει να το πετύχετε αυτό. Θέσατε επίσης και ένα ερώτημα για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Νομίζω ότι θα υπάρξει εδώ μια δυνατότητα να υπάρξει μια γνωμοδότηση και από τη δική σας Επιτροπή. Ξέρετε ότι οι επίτροποι έχουν συζητήσει πολλές φορές για τα ζητήματα αυτά που έχουν να κάνουν με τα γλωσσικά θέματα, τα οποία είναι πολύ δύσκολα. Θα έχουμε μία άτυπη συνάντηση το Σεπτέμβριο και μια πιο επίσημη τον Οκτώβριο. Εγώ θα προσπαθήσω να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση για τα θέματα αυτά. Δεν πρέπει να σας αποκρύψω όμως ότι οι συνθήκες προβλέπουν μια σειρά από εργαλεία για τα θέματα αυτά και για μένα η πρόθεση και η φιλοδοξία της Ευρώπης θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία στο επίσημο Συμβουλίο του Δεκεμβρίου. Γιατί τα θέματα αυτά που έχουν μείνει ακίνητα σε μεγάλο βαθμό εκκρεμούν ακόμα περίπου από τη δεκαετία του 1950. Αν θέλει λοιπόν η Ευρώπη να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να προχωρήσει σε μια πραγματιστική λύση, αυτό θα είναι θετικό και δεν σας κρύβω ότι η πρόταση του κύριου Μπαρνιέ η οποία έχει σαν στόχο να μειώσει το κόστος μετάφρασης για ένα δίπλωμα ευαισθητεχνίας από 12.000 ευρώ σε 700 και μόνο ευρώ, αυτό είναι κάτι το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις μας, ιδίως τις μικρομεσαίες. Για τη στοχευμένη εναρμόνιση που αναφέρατε, Νομίζω ότι έχω απαντήσει. Και τώρα, σε σχέση με το θέμα που αναφέρατε, με την έκθεση Μόντι και πώς θα υλοποιηθούν αυτά σε πιο συγκεκριμένες δράσεις, εγώ νομίζω ότι πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη τις προτάσεις που θα προέλθουν από τον Επίτροπο Μπαρνιέ, οι οποίες θα παρουσιαστούν το φθινόπωρο, και η έκθεση Γκρέχ και η συνεργασία η οποία έχει γίνει μέσα στα πλαίσια της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς είναι μεγάλη σημασία. Εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι με τις εκδηλώσεις που θα οργανώσουμε και ανέφερα ορισμένες προηγουμένως και μίλησε επίσης και ο πρόεδρος σας, ελπίζουμε ότι με τις εκδηλώσεις αυτές και με τις ε, επαφές αυτές θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε σημαντικό βαθμό. Η ιστορία της Ευρώπης θα πρέπει να είναι η ιστορία των πολιτών, των επιχειρήσεων, των καταναλωτών για να έχουμε μία ισορροπία και μία συνένεση να βλέπουν επίσης οι πολίτες μας ότι υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα τα οποία γίνονται προς τα εμπρός και αυτό πρέπει να το κάνει και η Βελική Προεδρία. Αυτά θα ήθελα να πω υπό μορφή απαντήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Ελπίζω ότι μπορείτε να μείνετε λίγο παραπάνω. 20 ε, λεπτά περίπου, ναι. Έξι συναδέλφους έχω ακόμη είναι δυνατόν να περιοριστείτε σε ένα περίπου λεπτό, κύριε και κύριοι συνάδελφοι. Θα σας δώσω, θα σας κάνω ένα νόημα για να σας ενθαρρύνω να τηρήσετε το ενα 15 λεπτό. Ε, ίσως υπήρξα υπερβολικά ανοιχτικός απέναντι στους πρώτους που ήταν όμως και οι εκπρόσωποι των κομμάτων. ας πούμε δύο λεπτά, επειδή είναι σημαντικές και οι προσωπικότητες του δεύτερου γύρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Υπουργό που είναι μαζί μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά. Αναφερθήκατε στον πρόεδρο Ντελόρ. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και σαν Γαλλίδα, διότι εδώ και 20 χρόνια λέω ότι το πνεύμα του Ντελόρ λείπει από την Ευρώπη και η Ευρώπη πεθαίνει. Ευχαριστώ πολύ που τον αναφέρετε. Λοιπόν, είσαστε στο Βέλγιο, εσείς ε, ε, υποδέχεστε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες που έρχονται να επισκεφθούν τους, ε, τα θεσμικά όργανα και ελπίζω ότι πραγματικά θα, θα συμπεριφερθείτε σαν πραγματικός Ευρω, και δεν θα διεκπαιρεώσετε τα θέματα όπως κάνουμε συνήθως. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία θέματα τα οποία αφορούν τους Ευρωπαίους πολίτες. Καταρχάς είναι το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Ε, όλοι και ο Επίτροπος Βαγνιέστο το και αν δεν ανήκω στο, στην πολιτική του ομάδα, είναι... Ε, έχουν απόψεις ε, που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Μιλάμε για... Ζούμε μια κρίση, ζούμε μια περίοδο κρίσης και όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε τους καταναλωτές. Δεύτερον, εσωτερική αγορά σαν ε, εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης ε, τα θέματα αυτά αφορούν τους καταναλωτές ε, αλλά και τους εκλεγμένους της τοπικής αυτοδιοίκησης διότι θα πρέπει όλοι, όλοι να συμμετέ... θέλουν να, στις δημόσιες αγορές να έχουμε συγκεκριμένα πρότυπα, δικλείδες ασφαλείας έτσι ώστε και οι, οι τοπικοί άρχοντες αν θέλετε να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα των κρατικών προμηθειών, των δημοσίων αγορών με διαφάνεια. Επίσης κάποιο άλλο θέμα το οποίο ξεκίνησε και επανεξεκίνησε μάλλον ε, η, Ισπανική Προεδρία για το δικαίωμα των ασθενών. Ε, ξέρω ότι το Βέλγιο έχει υγειονομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας ε, γίνεται μια συζήτηση και σε νομικό επίπεδο για την νομική προστασία αυτών των ασθενών που εποφελούνται από τις διασυνοριακές υπηρεσίες. Ήθελα να ξέρω εσείς πότε θα ξεκινήσετε ξανά τη συζήτηση και κατά δεύτερον θα λάβετε υπόψη ε, αυτό το οποίο θέλουν οι σοσιαλδημοκράτες, δηλαδή να μην έχουμε υγεία δύο ταχυτήτων και επίσης η υγεία να μην αποτελεί ένα καταναλωτικό αγαθό αλλά ένα αγαθό, έτσι ώστε να γίνει και αγαπητή η Ευρώπη. Ο καθηγητής Κρέντε Κάμπος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και την παρουσίασή σας εδώ. Είμαι πολύ ικανοποιημένο για την ε, αντιμετώπιση που έχετε έναντι του Κοινοβουλίου και τη συνενετική προσέγγιση που δείχνεται σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμφωνούμε όλοι για τη στρατηγική σημασία που επέχει η έκθεση Μόντι και την ανάγκη να υπάρξει μια ανάκαμψη της εσωτερικής αγοράς. Μπορεί να διαφέρουμε ίσως σε λεπτομέρειες, αλλά ακόμα και έτσι αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ μας. Εγώ συμφωνώ μαζί σας με αυτά που λέτε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια εσωτερική ψηφιακή αγορά, το ηλεκτρονικό εμπόριο με απλά λόγια, και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μην παραγνωρίσουμε, να μην ξεχάσουμε τις υπηρεσίες κοινοφελούς χαρακτήρα, είτε είναι δημόσιου χαρακτήρα ή γενικού οικονομικού συμφέροντος. Σήμερα βλέπουμε τα πράγματα καλύτερα από ό,τι πριν από δύο χρόνια. Είναι, είναι βέβαια ένα θέμα που έχει ιδεολογικές πτυχές, έχετε δίκιο, αλλά είναι απαραίτητο να έχουμε και μια διαυγή αντιμετώπιση για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα να σας θέσω δύο ερωτήματα σε σχέση με τις προθέσεις σας σε ό,τι αφορά την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Κάποια στιγμή η Κομισιόν μας παρουσίασε μια πρόταση ρύθμισης η οποία ουσιαστικά αποχωρίζει την πλήρη εναρμόνιση από την μερική εναρμόνιση, λέγοντας ότι τα συμβόλαια τα οποία δεν είναι πρόσωπο με πρόσωπο, δηλαδή τα ηλεκτρονικά συμβόλαια, θα πρέπει να έχουν μια ειδική ρύθμιση για να προωθηθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ τα συμβόλαια τα κανονικά, οι κανονικές συμβάσεις θα έχουν άλλη μεταχείριση. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η δική σας στάση ως Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητος. Δεύτερον, αναφερθήκατε ότι ένα μέρος της οδηγίας ένα μέρος τη ευθύνη μάλλον για αυτήν την οδηγία θα πρέπει να μείνει στην επόμενη Προεδρία. Εγώ θα ήθελα να είστε πιο σαφεί για το μέχρι πού θέλετε να φτάσετε στα πλαίσια αυτής της οδηγίας. Ευχαριστώ. Η κυρία Βάιλερ τέλος. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ με, με τη σειρά μου που θυμήσατε το πνεύμα των πράξεων του Ζακ Τελόρ για μένα ως Γερμανίδα σοσιαλδημοκράτησα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό να συμβαίνει αυτό. Θα μιλήσω κι εγώ πάλι για τις καθυστερήσεις πληρωμών ως εισηγήτρια με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να μην αναβληθεί ξανά και ξανά από το Συμβούλιο. Είπατε ότι πρόκειται για προτεραιότητα της Προεδρίας σας. Επενέσατε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την συμβαστική λύση που επιλέξαμε στην αποφάσισή μας. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία, αλλά το πράγμα είναι επίγον. Δεν είναι μονάχα οι εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμότητες, εκκρεμείς πληρωμές, είναι και οι χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις οι οποίες είναι αναγκασμένες να κατευθυνθούν στην πτώχευση διότι δεν πληρώνονται, δεν λαμβάνουν τα όσα τους οφείλονται. Κατ' επανάληψη έχει δεχθεί ότι ειδικά για να μην ανοίξει στο Συμβούλιο η πόρτα σε τόσες πολλές εξαιρέσεις, εγώ περιορίστηκα σε μια εξαίρεση και μόνη. Δεν θα περιλάβουμε τον κάθε παιδικό σταθμό και την ε, και το κάθε μικρό ίδρυμα, αλλά τα μεγάλα νοσοκομεία. Διότι τα νοσοκομεία στι περιφέρειες όπου λειτουργούν είναι και σημαντικοί οικονομικοί παράγοντε. Και όσο δημοκράτησα δεν θέλω καθόλου να χαίρουν προνομίων τα ιδιωτικά νοσοκομεία απέναντι στα κοινοτικά ή κρατικά. Νομίζω ότι αυτή η εξαίρεση πρέπει να παραμείνει. Εάν συμφωνήσει το Συμβούλιο θα βρει βεβαίω και σωστά επιχειρήματα. Αυτό είναι σημαντικό. Οι άλλε συμβαστικέ λύσει μετά από μακρές συζητήσεις εδώ στην Επιτροπή μας στο Κοινοβούλιο, εγκρίθηκαν με μεγάλη συνένεση, νομίζω με έξι μόνον αποχές. Σας προσφέρουν λοιπόν μια σοβαρότατη βάση και από τη σκοπιά των διαφόρων χωρών μελών, διότι συμμετέσχουν και χώρες του Νότου και του Βορρά και της Ανατολής και της Δύσης. Δεν ήταν μονάχα οι δύο μεγάλες χώρες μέλη, αλλά υπήρξε συνένεση διακομματικά και από, μεγάλες, και πολλές μάλλον χώρες Νομίζω λοιπόν θα σας προσφέρουμε μια πολύ στέρεα βάση. Δεύτερον, είπατε οι βελικές κυβερνήσεις συχνά έχουν αντιμετωπίσει θύελες αλλά έχετε ένα, στο Βέλγιο πάντως σίγουρα ένα καλό σύστημα κοινωνικών εξισορροπήσεων για τις ε, οδηγίες αναθέσεως συμβάσεων κλπ. Αν ληφθούν υπόψη και τα κοινωνικά κριτήρια, αυτό θα βρει σύμφωνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στα χαρτιά, στην οδηγία δηλαδή, υπάρχουν αυτά ήδη. Το ερώτημα είναι εάν όντως μπορεί να εφαρμοστεί με τον τρόπο αυτό στις χώρες μέλη. Και είπατε, μιλήσατε και για καινοτομία. Εγώ το βρίσκω ενδιαφέρον αυτό. Ένα καινοτόμο μέτρο θα ήταν εάν μπορούσαμε να συναντηθούμε με την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή του Βελγικού Κοινοβουλίου για να δούμε πώς εφαρμόζεται το δίκαιο εδώ της ανάθεσης συμβάσεων. Εντάξει, αν θέλετε απαντήσετε σε αυτούς και θα έχουμε και τους τελευταίους τρεις ομιλητές μετά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους για τις ερωτήσεις. Καταρχήν, Αναφερθήκατε κυρία μου στο Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Τεχνίας. Νομίζω ότι εδώ απήντησα αναφερόμενος σε αυτά που είπε ο κύριος Ροσφόρ. Τόνισα τη σημασία που εγώ αποδίδω στο σύστημα αυτό, το οποίο είναι απαραίτητο. Αλλά θέσατε και θέματα σε σχέση με τις δημόσιες προμήθειες και τα δικαιώματα των ασθενών. Για τις δημόσιες προμήθειες, όπως σας είπα, <clears throat> πιστεύω ότι το να θεωρούμε την ε, τιμή την προσφορά, τιμή προσφοράς ως μόνο κριτήριο εμποδίζει την καινοτομία και δεν λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια τα οποία αναφέρεται και στη Σύρια. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έρθει με μια πρωτοβουλία ε, ναυαρχίδα, η πρωτοβουλία Φάρο, μέσα στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Ευρώπη 2020 και μέσα στα πλαίσια αυτά με διαβεβαίωση η Κομισιόν ότι και τα θέματα των δημοσίων προμηθειών θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο και θα συμπεριλάβουν <clears throat> και τα κριτήρια που αναφέρατε εσείς, δηλαδή τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ε, άλλα κριτήρια. Ο στόχος εδώ είναι να εξασφαλίσουμε όμως και μία ασφάλεια δικαίου. Εγώ υπήρξα δημοτικός σύμβουλος και ξέρω πόσο μεγάλε είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όταν έχουμε να κάνουμε <clears throat> με δημόσιες προμήθειε. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε μια καλή εργασία για τα θέματα αυτά. Για τα θέματα υγειονομικής περίθαλψης. Οι υγειονομικές υπηρεσίε προφανώς δεν είναι ένα εμπορεύσιμο αγαθό και μόνο όπως τα άλλα αγαθά. Γι' αυτό είχαμε πολλές συζητήσεις στο Συμβούλιο για τα ζητήματα αυτά και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι πεπισμένος ότι οι συνάδελφοι από τα κράτη-μέλη γνωρίζουν ακριβώς αυτή την προβληματική και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο αυτή την προβληματική στο μέλλον <clears throat> και έχουμε φυσικά την, την εμπειρία του Βελγίου όπου ήδη υπάρχει κάποιο έργο το οποίο, κάποια εργασία που πρέπει να ολοκληρωθεί και βλέπουμε την ε, ιδιαιτερότητα αυτών των τομέων. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει μια συζήτηση και να επέλθουν κάποιες συμφωνίες και κάποιες λύσεις. Για τον ε, καθηγητή Κορέα Κάμπους, αναφερθήκατε στο θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Εγώ σας είπα ότι διάβασα με προσοχή την έκθεση Μόντι που αναφέρεται στην Ευρώπη του 2020. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια ενοποιημένη ηλεκτρονική αγορά στην Ευρώπη και θεωρούμε ότι ένα 4% του ΑΕΠ θα είναι αυτό το οποίο χρειάζεται για να εξασφαλιστεί η δημιουργία πλούτου στον τομέα αυτό του ηλεκτρονικού εμπορίου. Επομένως, ένα σημαντικό εγχείρημα. Αν συγκρίνουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη με αυτό που υπάρχει στις ΗΠΑ και σε άλλα μέρη του κόσμου, ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν προσκόμματα. και τα προσκόμματα, τα εμπόδια προέρχονται κυρίως από τις δυνατότητες πληρωμών. Αυτά εμποδίζουν την χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου από τους καταναλωτές. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια δικαίου για τους εμπόρους, αφενός, για να μπορεί να λειτουργεί καλύτερα το ηλεκτρονικό εμπόριο. Στη, στο νομοθέτημα για την ενιαία αγορά θα πρέπει <clears throat> να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Η Επίτροπος Κρούζ, η οποία είναι υπεύθυνη για την ψηφιακή ατζέντα, παρουσίασε σήμερα μία κέρια πρωτοβουλία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Καθηγητά, επίσης αναφερθήκατε στην διαφορά η οποία υπάρχει μεταξύ των, ε, <clears throat> της χρήσης των υπηρεσιών επιτοπίως ή εν κινήσει σε, άλλες, ε, σε άλλους χώρους. Η κυρία Ρέντινγκ λοιπόν <clears throat> στην περίπτωση αυτή θέλει να κάνει αυτή τη διαφοροποίηση μεταξύ on-premises και off-premises όπως αναφέρεται και αυτά θα ε, Όλα αυτά εξετάστηκαν ήδη από την Ισπανική Προεδρία. Και υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες έχουν καταφέρει να προχωρήσουν σε μια τέτοια διαφοροποίηση. Αλλά πολλές οργανώσεις επαγγελματικές θεωρούν ότι μια τέτοια διάκριση δεν μπορεί να διατηρηθεί με ευκολία. Γι' αυτό δεν μου φαίνεται μια ιδιαίτερα βιώσιμη λύση. Κυρία Βάιλερ, επίσης, κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών παρατηρήσεων, εγώ Αναφέρθηκα ηθελημένα στην εκθεσή σας. Ξέρω ότι έχετε κάνει πολλά πράγματα στην κατεύθυνση αυτή. Και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι εάν θέλουμε να βρούμε μια λύση για τις καθυστερήσεις πληρωμών, από τη στιγμή που θα έχει ξεπεραστεί η χρηματοοικονομική κρίση, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το εξή παράδοξο. Έχουμε την κρίση. Πρέπει να βρούμε μια λύση για την κρίση. Και αυτό το θέμα έχει μείνει ανοιχτό για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά θα πρέπει να συμβιβάσουμε αντιμαχόμενα συμφέροντα στο σημείο αυτό. Σα υπενθυμίσω αυτό που είπε ο κ. Σουάμπ για τι επαφέ business to business. Νομίζω ότι πολλοί θεώρησαν ότι μπορούσαμε να βρούμε εκεί μια συμβαστική λύση. Αλλά αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία παραπέμπονται στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων για να προσπαθήσουμε να δούμε αν υπάρχει έδαφος για να υπάρξει μια κοινή θέση και μια εντολή για να μπορέσει να βρεθεί μια κοινή λύση για όλα αυτά τα θέματα. Και για μένα είναι από τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Βελική Προεδρία. Ίσως ακόμα και αυτή τη βδομάδα στην Κορεπέ θα μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό. Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα αυτό. και νομίζω μπορούμε να βρούμε μια λύση με όλους τους εμπλεκόμενους στην Ευρώπη. Αναφερθήκατε λοιπόν <clears throat> επίσης και σε κάποιο άλλο θέμα για το οποίο θέλω να σας πω ότι εμείς προσκαλέσαμε την Επιτροπή σας να έρθει σε επαφή με τις δικές μας υπηρεσίες Βρυξέλλες για να σας δείξουμε πώς λειτουργεί το θέμα αυτό, πώς προσπαθούμε να επιτύχουμε την υλοποίηση, την πρακτική υλοποίηση αυτών των ε, ρυθμίσεων και θα πρέπει ακόμα να συνεργαστούμε με τον πρόεδρο της Επιτροπής σας για να οργανώσουμε αυτή την επίσκεψη, αλλά νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα από μία από τις επαφές που θα οργανώσουμε κατά τη διάρκεια της ε, προεδρίας μας. Ας έρθουμε στους τελευταίους ερωτώντες κυρία Κορατσπέλτς, κυρία Τάιλερ, που είναι και η συγγήτρια για τα οικοδομικά ειδικά, και η κυρία Ράπτη. Θα παρακαλέσω και πάλι να αρκεστείτε σε δύο λεπτά οι ερωτώσεις και οι ερωτώντες. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Συγχαίρω και εγώ, σας συγχαίρω και εγώ και σας ε, ευχαριστώ κυρίως για την αιμονή σας στην κοινωτική προσέγγιση. Τώρα, για την οδηγία για την προστασία καταναλωτών. Ναι, μεν το Κοινοβούλιο προ δύο εβδομάδων ενέκρινε τη διαγραφή των κεφαλαίων 6 και 7 στην ε, οδηγία προστασία των καταναλωτών για την επισήμανση των τροφίμων με ετικέτες κλπ. Μιλούμε για αγορά των καταναλωτών. Χειροκροτούμε την έκθεση Μόντι που μιλεί για μια ενιαία αγορά. Αλλά όταν παρακολουθήσετε την ε, ε, συζήτηση θα δείτε ότι είναι ή η αγορά ή οι καταναλωτές. Γιατί η νομοθεσία γιατι την νομοθεσια προστατευει τις επιχειρήσεις. Απευθύνω έκκληση λοιπόν, αλλά ε, ζητώ και τις απόψεις σας για το πώς μπορούμε να επαναφέρουμε το όραμα ότι η εναρμόνιση, οι κοινοί κανόνες, η κοινή αγορά είναι εποφελής και για τους καταναλωτές, δηλαδή με ασφάλεια δικαίου, με διαφάνεια που να είναι εποφελής όπως είπα για τους καταναλωτές. Ποιο, θα πληρώσει το τίμημα μια ενιαία νομοθεσία έτσι 27 διαφορετικέ. Ορισμένα κεφάλαια θα είναι πλήρω εναρμονισμένα, άλλα θα είναι εν μέρη εναρμονισμένα και ούτω καθεξής. Ο εισηγητή μα έχει κάνει μια εξαιρετική εργασία και εγώ θα τον αποκαλώ καβούρα από εδώ και μπρο. Όποιο γνωρίζει τελική ιστορία θα καταλάβει γιατί. Για να βάλουμε ένα στόχο για την εναρμόνιση, παρόλα αυτά υπάρχει ακόμη ανάγκη πολιτικού οράματος που ελπίζω να μπορέσετε να εμπνεύσετε στο Συμβουλίο, ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από, ε, μια, από ένα εγχείρημα συγκριτικού δικαίου και να φτάσουμε ξανά στην υλοποίηση του πνεύματος της ενέας αγοράς που θα είναι αμοιβαία υποφελής και για τον καταναλωτή και για την επιχείρηση. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ κύριε Μπίλτ. Κύριε Τάιλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ζητώ συγγνώμη για την ε, καθυστέρησή μου, αλλά συζητούσα για θέματα οικοδομικών υλικών. Χαίρομαι για το ανοιχτό πνεύμα που δείχνετε. Χαίρομαι που αναφερθήκατε και στην οδηγία για τα οικοδομικά υλικά. Εγώ θα συναντηθώ με τους και συνεισηγητές μου αύριο. Λίγα τώρα σχόλια σύντομα. Πρώτα, για ένα θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο για την πώληση εξ Εάν δεν σέβεται τους κανόνες μια μεγάλη επιχείρηση, υπάρχει μέγα κίνδυνο να, το, να ακολουθήσει το παράδειγμα του και άλλοι. Υπάρχει μια υπόθεση. Μπορείτε να μας πείτε τα γνώμη σας δεύτερον τώρα για ε, κρυφά, κρυμμένα μάλλον, ε, έξοδα πιστοτικών καρτών. Πολλοί που πηγαίνουν τώρα στις ε, διακοπές το ίδιο ισχύει και για τα κινητά τηλέφωνα και πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν τώρα στι διακοπέ και αρχίζουν ήδη από 1η Ιουλίου οι μετακινήσει αυτέ. Άνθρωποι που χρησιμοποιούν τα κινητά του τηλέφωνα και στην Αλοδαπή και ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι έχουν να πληρώσουν πολύ περισσότερα όταν επιστρέφουν. Αυτά ανισχύουν πολύ τον κόσμο. Μίλησαμε και για την πολιτική καινοτομία. Γνωρίζω ότι θα υπάρξει πρόταση τον Σεπτέμβριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι συνάδελφοί μα τη Επιτροπή Βιομηχανία ενδιαφέρονται ιδιαίτερα. Η καινοτομία όμω ενδιαφέρει και εμά. Έχετε κάνει κάποιες σκέψεις από αυτού. Μου αρέσει και πολύ ο τίτλος σας για αυτό το streamlining που έχετε ε, στον τίτλο σας ως υπουργό. Ποτέ δεν έχω ξανακούσει για υπουργό αρμόδιο για streamlining. Βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και σας εύχομαι να έχετε καλή επιτυχία στην εργασία σας. Ωραία κυρία Τάριερ. Η ε, κυρία Ράπτη παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου και εύχομαι κάθε επιτυχία στη δουλειά σας. Ε, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν είδατε αυτό το newsletter που βγαίνει με πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ χρήσιμο και κυρίως έχει πάρα πολύ καθαρές φωτογραφίες. Στη φωτογραφία που μας περιγράψατε εσείς για την εσωτερική αγορά, εγώ δεν μπορώ να διακρίνω καθαρά τους πολίτες, δηλαδή τους καταναλωτές. Και αυτό μου δημιουργεί σκέψεις. Όπως περισσότερες σκέψεις μου δημιούργησε και η απάντηση που δώσατε στην ερώτηση της συναδέλφου μου Μπερναντέτα για τις υγειονομικές υπηρεσίες. Στις υγειονομικές υπηρεσίες κυρίως συναντούμε πολίτες, καταναλωτές και μάλιστα ασθενείς. Ε, νομίζω ότι μας δώσατε ως απάντηση και σε αυτό το σημείο ένα πολύ ωραίο πακέτο με ένα πολύ ωραίο αμπαλάζ, αλλά έχω ερωτηματικά για το περιεχόμενο. Θέλω να ευχηθώ και πάλι καλή επιτυχία στη δουλειά σας και να ακούσω τις σκέψεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ράπτη και σας ευχαριστώ που επενέσατε το newsletter. Αν μας στείλετε email θα σας στείλουμε το newsletter αυτό και θα σας το στέλνουμε τακτικά ε, προσωπική, προσωπικό αντίγραφο να έχετε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ. Μπορώ να μιλήσω αγγλικά. Ωραία, το πνεύμα της ενιαίας αγοράς. Σωστό. Έχουμε 27 ή 28 διαφορετικά καθεστώτα. Μπορούμε να δούμε ποια είναι τα καλύτερα, να, να, βρούμε δηλαδή ε, να κάνουμε αυτό το cherry picking. Ε, εγώ ως αρμόδιος υπουργός ή μάλλον να το πω διαφορετικά, αν θέλει κανείς να δημιουργήσει μια ενιαία αγορά βασισμένη στην οδηγία προστασίας καταναλωτών. Αυτό που χρειάζεται κανείς είναι μια νέα ισορροπία, μια πραγματική ευρωπαϊκή ισορροπία. Μια εξισορρόπηση δηλαδή ανάμεσα στα συμφέροντα των καταναλωτών και των επιχειρηματιών. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι δυνατόν. Αυτό που χρειάζεται κανείς είναι πολιτική που δεν θα υπερασπιστούν μόνο τα συμφέροντα της χώρας μέλους τους, αλλά που θα επιζητήσουν την δημιουργία μια, μιας αγοράς η οποία να είναι πιο δυναμική. Χρειάζεται πιο πολύ δυναμισμό η, η Ευρώπη. Χρειάζεται αυτή την διάθεση των επιχειρήσεων ε, να δραστηριοποιηθούν και πέραν των συνόρων, προσφέροντα υπηρεσίε και αγαθά στου καταναλωτέ. Όπω απάντησε και στον καθηγητή προηγουμένω, το ηλεκτρονικό εμπόριο Εφόσον όμως δεν προσφέρει την ε, ασφάλεια δικαίου στους καταναλωτές, ότι δηλαδή τα δικαιώματά τους θα, ε, τα συμφέροντά τους θα ε, προστατευτούν επαρκώς, δεν έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει η ευρωπαϊκή θεώρηση να είναι μέσα στα πλαίσια, μέσα σε αυτό το πνεύμα. Το ότι αναφέρθηκα στον Ζακ δεν έχει σχέση με το ότι είναι Γάλλος και ευφύ άνθρωπος, αλλά ότι πραγματικά προσωποποίησε, προσωπι, προσωποποιούσε, δηλαδή στο πρόσωπό του, αν θέλετε έτσι, υλοποιούνταν αυτό το πνεύμα της ενιαίας αγοράς. Και μακάρι να υπήρχε περισσότερος Delors τώρα. Υπάρχει ακόμα το πνεύμα αυτό της ενιαίας αγοράς. Και από την σκοπιά των προεδριών, όταν μιλούμε με τις χώρες μέλη και ε, ε, προσπαθούμε να τις πείσουμε ότι χρειάζεται μια νέα βάση. Κύριε Τάιλερ, κύριε Τάιλερ μιλήσατε για το πακέτο των, ταξιδιών. Το 2011 θα υπάρξει σχετική πρωτοβουλία από την Κομισιόν, υπό Ουγγρική Προεδρία επομένω. Και για την καινοτομία, μιλήσατε για αυτή την ε, πρωτοβουλία Φάρο. Εγώ αναφέρθηκα στην πρωτοβουλία Φάρο επίσης, γιατί είχα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον αρμόδιο επίτροπο για καινοτομία και αυτό που νομίζω ότι απαιτείται ε, για την καινοτομία είναι μέσα στα πλαίσια αρμοδιοτήτων που έχει η Ευρωπαϊκή ε, ε, Ένωση για εναρμόνιση των προδιαγραφών για τις δημόσιες προμήθειες. Εκεί χρειάζεται να γίνει κάποια πρόοδος αυτό θα προσπαθήσω να επιτύχω και ελπίζω να μπορέσουμε να επιτύχουμε αποτελέσματα. Αναφερθήκατε σε μια συγκεκριμένη υπόθεση, την υπόθεση NEX. Πρόκειται για ένα παράδειγμα που δείχνει ότι δεν απαιτούνται μονάχα οι κανόνες, αλλά και η ε, ενεργός δραστηριοποίηση των εθνικών εποπτικών αρχών. Δεν ξέρω αν ήσασταν παρούσα εκείνη τη στιγμή. Το, μίλησα ότι θα έχουμε ε, τις ε, ε, inspection days και το, Σεπτέμβριο του 2010 με προσκλήσεις και προς επιχειρήσεις από άλλες χώρες μέλη για ε, την ε, συμμετοχή τους. Αν έχουμε καλή συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών, αυτή θα αποδώσει. Αλλά βέβαια χρειάζονται κοινοί κανόνες και αυτό είναι σημαντικό να επιτευχθεί για την προστασία των καταναλωτών. Για την κυρία Ράπτη, αναφερθήκατε στους ασθενείς και αναρωτηθήκατε τι υπάρχει μέσα στο πακέτο. Στο φόρουμ ενίας αγοράς που θα οργανωθεί στις 9 Νοεμβρίου χάρη και στις προσπάθειες της δικής σας Επιτροπής θα αφιερωθεί χρόνος και ενέργεια στη συζήτηση αυτού του θέματος των ασθενών και στην αναγκαιότητα να βρεθούν λύσεις υπέρ αυτών. Όταν αναφέρθηκα στα όσα είπε η κυρία σας Μπερναντέτ για τα συστήματα υγείας, το έκανα αυτό διότι γνωρίζω τις ευαισθησίες που περιστρέφονται γύρω από αυτό το θέμα και νομίζω ότι και εκεί οφείλουμε να επιτύχουμε κάποιο βαθμό συνεργασίας μεταξύ χωρών μελών. Νομίζω ότι ε, διαθέτοντας χρόνο, εγώ θα είμαι παρόν στις 9 Νοεμβρίου, διαθέτοντας χρόνο λοιπόν για τη συζήτηση αυτή, νομίζω θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις που μου έθεσαν οι συναδελφοί σας. Είναι πραγματικά μια σημαντική πρόκληση για μένα να ε, καλούμε να απαντήσω σε ερωτήσεις ανθρώπων που έχουν σημαντικό ενδιαφέρον για αυτά τα θέματα στην αρχή της Προεδρίας μας. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία αυτή να καταστήσω γνωστές τις θέσεις μου. Θα συνεργαστούμε στη διάρκεια των προσεχών εξημινών της Βελικής Προεδρίας όπου θα συμμετάσχω και εγώ σε αυτό τον ευρωπαϊκό χώρο και ελπίζω ότι στο τέλος των 6 θα μπορέσουμε να σημειώσουμε κάποια σημαντικά αποτελέσματα μια θετική συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την καταπληκτική αυτή επίδοσή σας στην κάλυψη όλων αυτών των τομέων. Πιστεύω ότι σίγουρα τα θέματα των δημοσίων προμηθειών μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και έχουμε φυσικά εδώ πέρα την έκθεση της κυρίας Ρίλε η οποία αφορά το θέμα αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για τις πολλές πρωτοβουλίες που παίρνετε και οι ημερομηνίες που αναφέρετε το Σεπτέμβριο θα είμαστε μεν στο Στρασβούργο και δεν θα μπορούμε να είμαστε παρόντες αλλά με μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε αυτή την εκδήλωση εξ αποστάσεως, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η εποπτεία της αγοράς και η ασφάλεια των καταναλωτών. Προσβλέπουμε λοιπόν στο να συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί σας και τους συνεργάτες σας και σας ε, ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο εξάμεινο της Βελικής Προεδρίας. Uh, Οπότε κυρίε και κύριοι, περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι η περίφημη οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Θα επιτρέψω να επανέλθετε όλοι στα έδρανά σας και αναμένουμε επίσης και την επιστροφή του εισηγητού ο οποίος έχει αποχωρήσει για ένα σύντομο διάστημα, είμαι σίγουρος ότι θα επανέλθει, να ελέγξω μονάχα ποιοι είναι οι σκιώδεις σήμερα. από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Η, Βανιούτ, η κυρία Βανιούτ, η κυρία Γκέπχατ, Ροσφό, Τούρουνεν. Ο κ. Μπίνεν δεν είναι παρόν. Ο κ. είναι εδώ. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε ένα πρώτο γύρο συζήτησης ή μάλλον σήμερα ένα πρώτο γύρο γιατί είναι τουλάχιστον τρίτη ανταλλαγή απόψεων που είχαμε και είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων την προηγούμενη φορά. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν και τον εισηγητή για την τόσο επικοδομητική συνάντηση που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα με όλους τους σκιώδεις εισηγητές και θα δώσω το λόγο και στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, Ίκοθεν Νοήτ. Δίνω λοιπόν το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Σουάμπ, να συνεχίσουμε να συνεχίσει τη συζήτηση για την έκθεσή του. Ευχαριστώ και Πρόεδρε. Μετά την ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον ε, Βέργο Υπουργό θα περιοριστώ σε σύντομα σχόλια ώστε να μπορέσει να γίνει και συζήτηση. Στην βάση της επισκόπησης που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ... λίγων εβδομάδων παρακάλεσα τους συνεργάτες μου να περιλάβουν και τα συμπεράσματα της εκθεσής μου τον πίνακα αυτό. Ακόμα όμως δεν είναι ολοκληρωμένη η εργασία αυτή. Δείχνει όμως ποιες μπορούν να είναι οι τροποποιήσεις της ε, οδηγίας εάν εγκριθούν οι τροποποιήσεις που προτείνω. Πρώτα ε, πάντως θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους που υπέβαλαν ε, προτάσεις, η κριτική, η έπαινο προς εμένα προσωπικά. Επίσης οι διάφορες οργανώσεις καταναλωτών ε, ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Δεν μπόρεσα να διαβάσω όλα τα σχόλια. Ε, συχνά είναι πολύ περίπλοκα τα θέματα, πάντως ε, υπόσχομαι σε όλες και όλους ότι θα απαντήσω προσωπικά και πλήρως. Τρίτο, μετά από την συνάντηση με τους πιο δυσηγητές την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν τεθεί ορισμένα θέματα τα οποία οφείλουμε να συζητήσουμε. Οι προτάσεις για τροποποίηση του εγγράφου της Κομισιόν κατέστησαν απαραίτητες διότι και στο Συμβούλιο αλλά και εδώ έχει ζητηθεί αυτό από τους συναδέλφους μου. Έχοντας υπόψη τις διάφορες συζητήσεις και ανταλλαγής απόψεων στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, έχω νομίζω μπορέσει να προσεγγίσω τα σημεία εκείνα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συνενέσεως και τα οποία θα είναι τα εξής. Πρώτον, χρειαζόμαστε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό πνεύμα ε, για την οδηγία αυτή. Αυτή η κόποση της ενιαίας αγοράς, την οποία επισημαίνει ο κ. Μόντι, δεν πρέπει έτσι απλά να την αποδεχθούμε. Χρειάζεται λοιπόν να προωθήσουμε μια πραγματική ενιαία αγορά καταναλωτικών αγαθών και από σκοπιανομική. Με τον τρόπο αυτό βέβαια δεν επιλύονται όλα τα προβλήματα της έννοιας αγοράς. Αυτό είναι σαφές, χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά. Αλλά πάντως θα αποτελέσει τουλάχιστον ένα βήμα. Άλλωστε οι τροποποίησεις που προτείνονται βασίζονται στην πεποίθηση ότι όλες αυτές οι αλλαγές πρέπει να οδηγήσουν σε μια καλύτερη συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων του καθενός. Για παράδειγμα και ο κανονισμός των δικαιωμάτων των επιβατών που θα το δει κανεί σε όλα τα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο μεταξύ ε, σημειώνουν όλοι ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν πλέον πολύ καλύτερα τα δικαιώματά τους, γνωρίζουν από ποιο λεπτό της καθυστερήσεως και μετά ε, μπορούν να τα απαιτήσουν και το καθεξής. Άλλωστε, όπως είπαμε και με τον Βέλγο Υπουργό, νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι θα υποσχεθούμε στους καταναλωτές ότι θα επωφεληθούν από την οδηγία δεν θα τους υποσχεθούμε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Θα τους υποσχεθούμε ότι εν τέλει θα προκύψει κάτι το οποίο θα είναι εποφελές για όλους τους καταναλωτές και καταναλώτριες αλλά και για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις. Στους τομείς εκείνους όπου ακόμη δεν έχει επιτευχθεί η συνενεσία αυτή διότι υπάρχουν διαφορετικές εθνικές παραδόσεις, γιατί υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις, γιατί υπάρχουν προβλήματα που δεν έχουν ακόμα επιληθεί. Η πρόταση προβλέπει την ελάχιστη εναρμόνιση ως εξαίρεση του άρθρου 4. Για παράδειγμα, για τις εγγυήσει, για την έναρξη των εγγύσεων, αλλά και για την αντιστροφή του βάρους αποδείξεως. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε 7 συγκεκριμένα σημεία για να εξηγήσω για ποιο λόγο φέρει δικαίως τον τίτλο της προστασίας των καταναλωτών. Έχουμε διευρύνει τις ε, συμβάσεις κατά την αξία τους. Με την κατάργηση του κατοφλίου εμπίπτουν πλέον όλες οι συμβάσεις στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Δεύτερο, για τις ε, πάλι για την εφαρμογή της οδηγίας έχει διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή ώστε να περιλαμβάνονται όλες οι επισκέψεις ε, των και περιλαμβάνονται επίσης και οι πρακτικές ορισμένων αεροπορικών επιχειρήσεων για παράδειγμα οι οποίες δεν ανακοινώνουν ε, εξ αρχής όλο όλα τα στοιχεία κόστους. Σε 12 εξάλλου χώρες μέλη οδηγούμε σε βελτίωση των προθεσμιών, οι οποίες είναι για την ώρα πάρα πολύ σύντομες. Αλλού τηρούνται, ε, τηρείται το status quo. Πέμπτο στοιχείο, εφόσον δεν εξηγούνται τα δικαιώματα των, ε, των καταναλωτών πριν από την σύναψη της συμβάσεως, πάλι εκεί προβλέπονται διαφορετικές προθεσμίες. Έκτο, σχετικά με, την, με τον κίνδυνο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Υπάρχει ωστόσο βελτίωση στην κατάσταση στην Ιταλία και στην Γαλλία και επίσης υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στην Ισπανία. Έβδομο, σχετικά με τα τετραγωνάκια στα οποία βάζει κανείς ένα σταυρό για τις ε, ε, συμβάσεις αυτές, στο μέλλον δεν θα είναι δυνατόν να ε, γίνονται ορισμένες παρερμηνίες και επομένως βελτιώνονται οι ε, διατάξεις υπέρ των καταναλωτών. Επίσης θα πρέπει ογδόν από εδώ και πέρα να είναι απόλυτα διαφανές το περιεχόμενο των γενικών συνθήκων που, ε, των γενικών όρων μάλλον ασκήσεως της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επομένως της συμβάσεως. Τώρα, όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε μια συνάντηση με τους πιο δυσηγητές και έχω μια ερώτηση για το θέμα του άρθρου 4 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το light motif της πρότασής μου είναι η στοχευμένη εναρμόνιση. Αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προβλέψει γενικά εναρμόνιση. Τώρα την έχει κάπως περιορίσει. Η βασική αρχή θα πρέπει να είναι εναρμόνιση, αλλά να υπάρχει και η ευκαμψία, η ευελιξία, να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Γι' αυτό θα ήθελα τώρα, ιδίω μετά από την συνάντησή μας της προηγούμενης εβδομάδας, να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θεωρεί ότι πρέπει να διατηρηθεί το υφιστάμενο σύστημα της ελάχιστης εναρμόνισης, ανεξαρτήτως του εάν θα θεωρηθεί απροσμίξτ ή αν θα θεωρηθεί ως leitmotiv. Και δεύτερο, αυτή η προσέγγιση της ελάχιστης εναρμόνισης συμβαδίζει με την νομική βάση του άρθρου 14 της συνθήκης. Κατά τη γνώμη μου, θα είναι συμβατό με την ε, ε, συνθήκη μόνο εάν υπάρξει γενικότερη εναρμόνιση και όχι μόνο μία απολύτως ελάχιστη εναρμόνιση. Η ερώτηση επίσης έχει το νόημα τι μπορεί, τι μπορεί να γίνει αν τροποποιηθεί η νομική βάση. Επίσης θα ήθελα να μάθω και τι θεωρούν οι συνάδελφοί μου σχετικά και για την βελτίωση της προστασίας άλλων δικαιωμάτων των καταναλωτών μέσω της αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε τον κύριο Μπρόγκ να, καταγράψει ερωτήσεις. Ε, θα πάρει το λόγο όμω αργότερα. Λοιπόν, α συνεχίσουμε τις συζητήσει, η κυρία Βάνιου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη γιατί εγώ δεν είμαι σκιώδη συγγήτρια όπως το ξέρουμε. Η κυρία Γκέπχαρτ είναι. Αλλά είναι απούσα. Ξέρω ότι ο κύριος Σβάμπ συνάντησε την προηγούμενη εβδομάδα τους σκιώδη συγγητέ και έγινε μια συζήτηση αρκετά ζωηρή θα έλεγα στην τελευταία συνάντηση της Επιτροπής ΙΝΚΟ. Πιστεύω ότι το βασικό, και αυτό δεν θα είναι εύκολο, θα χρειαστεί χρόνος, είναι να βρούμε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα σε μια ελάχιστη εναρμόνιση, η οποία είναι απαραίτητη, γιατί μέγιστη εναρμόνιση δεν μπορεί να γίνει, γιατί θα κατέβουν τα στάνταρ για τους καταναλωτές σε πολλές χώρες, αλλά τέλος πάντων ε, είναι μέγιστη και την ελάχιστη εναρμόνιση με κάποιες εξαιρέσεις. Το πρόβλημα είναι όμως ποιες θα τις εξαιρέσεις και ποια θα είναι η ισορροπία. Υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά το δίκαιο των συμβάσεων. Ε, εκεί θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Αυτό θα πρέπει να το προσπαθήσουμε και εκεί θα πρέπει να δείξουμε ένα ευρωπαϊκό πνεύμα, σαν και αυτό που ανέφερε και ο Υπουργός προηγουμένως. Η πλήρη και η στοχευμένη εναρμόνιση φαίνεται ότι είναι συγκρουόμενες έννοιες. Δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εναρμόνιση ε, και να είναι στοχευμένη. Αν είναι πλήρης εναρμόνιση θα μας πάρει πολύ καιρό ή θα πρέπει να έχουμε μια στοχευμένη εναρμόνιση ε, σε κάποιες χώρες για κάποιους τομείς ξέρω ότι το έχετε ζητήσει με την Εύλην και καταλήξατε σε κάποια συμφωνία, αλλά θα ήθελα να μας επιβεβαιώσετε το νέο χρονοδιάγραμμα, το οποίο φαίνεται να είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο αναφέρεται σε αυτή την επιστολή. Αυτό που αναφέρεται σε επιστολή είναι λίγο πιεστικό. Ξέρω ότι στις διακοπές θα σκεφτούμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες, τις οδηγίες που είναι ουσιαστικές, αλλά χρειαζόμαστε χρόνο. Ε, το χρονοδιάγραμμα που προβλέπετε μας οδηγεί λίγο προς το τέλος του 2010, αν κατάλαβα καλά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ροσφόρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη νέα εικόνα την οποία μας παρουσίασες. Δεν μπορώ να την ε, χωνέψω αν θέλετε αμέσως, να την ε, οικειοποιηθώ, αλλά η πρώτη ιδέα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι ε, ακόμα δεν μπορώ να την, δεν μπορώ να την αξιολογήσω. Και υπάρχουν πολλές αλλαγές ε, και για πολλές χώρες και για πολλά άρθρα πάρα πολλά πράγματα αλλάζουν και όπως ξέρετε πολύ καλά σε κάποια ε, κατάσταση άγχους που επικρατεί λόγω της οικονομικής κρίσης ε, και της δυσπιστίας απέναντι στην εσωτερική αγορά οι καταναλωτές δεν χρειάζονται πολλές αλλαγές σε, όσον αφορά το νομικό πλαίσιο και δεν ξέρω και αν οι επιχειρήσεις πιστέλουν. Τέλος πάντων η ουσία είναι ότι γίνονται αλλαγές και το βασικό για μένα δεν είναι να δούμε κατά πόσον αλλά οι θετικές αλλαγές είναι περισσότερες από τις αρνητικές. Δεν θα κάνουμε μια ισορροπία, δεν θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε μια ισορροπία ανάμεσα στις βελτιώσεις ή στις ε, επιδεινώσεις αν θέλετε της κατάστασης. Το πρόβλημα είναι αν επιδεινώνεται η κατάσταση αυτή η επιδείνωση είναι αποδεκτή ή όχι. Και οι αλλαγές αυτές μπορούν να δημιουργήσουν μια αίσθηση καχυποψίας στην αγορά ή δυσπιστία στην αγορά. Και για, να σας, ε, και για να αναφερθώ και στην γαλλική πραγματικότητα, υπάρχουν, πιστεύω, κάποια δικαιώματα των καταναλωτών, τα οποία ισχύουν μεν, αλλά δεν εφαρμόζονται δε. Άρα θα πρέπει να δούμε και τι ακριβώς ισχύει και, όχι, και τι εφαρμόζεται και όχι μονάχα το θεωρητικό επίπεδο. Τα επόμενα χρόνια πιστεύω ότι θα συζητηθούν πάρα πολλά ε, πάνω σε αυτό το θέμα σε όλες τις χώρες και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι δύο συμπληρωματικέ παρατηρήσει και βέβαια μετά θα πρέπει να συνεχίσουμε τι συζητήσει ε, και θα πρέπει και οι συνάδελφοι που δεν είναι σκιώδεις ηγητέ να πάρουν το λόγο μια και έχουμε τη δυνατότητα να εργαζόμαστε ε, σε τακτική βάση. Υπάρχει το άρθρο 4. Και όντω θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το θέμα και να δούμε πόσο θα το δούμε με το, με το Συμβούλιο. Ίσως να ψάχνω τη φιλοσοφική λίθο για το άρθρο 4 και επειδή είμαι αρκετά λογικός, δεν νομίζω ότι θα βρούμε την φιλοσοφική λίθο εδώ. Αλλά τέλος πάντων, επί της ουσίας, το άρθρο 4 δεν σημαίνει ότι όταν έχουμε ελάχιστη εναρμόνιση τα πράγματα είναι χειρότερα από ότι αν είχαμε μία μέγιστη εναρμόνιση. Εγώ θα ήθελα το άρθρο 4 να μας οδηγεί σε κάποια ισορροπία και συντακτικά το καταφέρνουμε τουλάχιστον. Διότι λέμε ότι η μέγιστη εναρμόνιση σε ορισμένε περιπτώσεις και ελάχιστη εναρμόνιση σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Όμως Δεν είναι σαν να λέμε ότι τώρα ε, προτιμάμε την λιγότερο κακή λύση και ότι ε, η λιγότερο κακή λύση είναι η εναρμόνιση, ενώ το καλύτερο θα ήταν η ελάχιστη εναρμόνιση, ενώ το καλύτερο θα ήταν η μέγιστη εναρμόνιση. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να καθαρίσουμε καταρχά τι θέλουμε και μετά θα δούμε πώ θα είναι η σύνταξη του άρθρου. Τώρα και κάτι άλλο το οποίο δεν αφορά το άρθρο 4, αλλά το οποίο επαναλαμβάνεται στο κείμενο, είναι το περίφημο τεστ αντοχής και συμβατότητας για τις εξαιρέσεις στα κράτη-μέλη. Εγώ θα ήθελα τα κράτη-μέλη προφανώς να κοινοποιούν στην Κομισιόν το κείμενο των εθνικών διατάξεων που παρεκκλίνει από το κείμενο εδώ, έτσι ώστε η ελάχιστη εναρμόνιση να γίνει με πλήρη διαφάνεια. Αντιμετωπίσω με ιδιαίτερο σκεπτικισμό τις λέξεις που χρησιμοποιούνται εδώ. Όταν λέμε ότι κάποιος είναι απολύτως απαραίτητο για την ε, προστασία του καταναλωτή, τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει απολύτως απαραίτητο ή απολύτως αναγκαίο. Και εάν βρούμε κάποιες λέξεις οι οποίες δεν είναι τόσο απόλυτες, ίσως η, το, η έννοια να αλλάζει. Αυτό το οποίο δεν θέλω όμως με τίποτα είναι τα κράτη να έχουν μια κοινοτική διαδικασία μένα, αλλά ε, καλούνται να εφαρμόσουν κάποιες, δια, κάποιες διατάξεις οι οποίες είναι τόσο άκαμπτες που σημαίνει αυτό ότι η εθνική τους νομοθεσία μετά δεν θα μπορέσει να εφαρμόσει. Δηλαδή, δεν θα εφαρμοστεί, συγγνώμη. Άρα, εάν υιοθετηθεί μια τέτοια διατύπωση, τι σημαίνει αυτό το απολύτω αναγκαίο, τι χρειάζεται απολύτω, τι είναι το απολύτω αναγκαίο για μια γυναίκα και έναν άντρα. Να ντύνεται, να τρώει, να εργάζεται κτλ. Αλλά το πρόβλημα είναι πώ μπορούμε να βρούμε κάτι το οποίο να μα καθησυχάζει και στο μέλλον. Τέλο πάντων, αυτά είχα να πω τώρα επί του παρόντο. Κατά τα λοιπά έχουμε και όλες αυτές τις τροπολογίες ε, οι οποίες θα μας απασχολήσουν. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη ποια είναι η, η, η λύση την οποία θα θετήσουμε καταρχάς για το άρθρο 4, για την διατύπωση και για το πόσο θα ε, διατυπώσουμε αυτό το, τη δοκιμασία συμβατότητας, θα δούμε και τι θα γίνει μετά ας πούμε σε περιπτώσεις διαφορών. Λοιπόν, ας ξεκαθαρίσουμε αυτά τα θέματα και μετά θα δούμε τι θα γίνει με τις τροπολογίες, πώς θα βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση. Κάτι το οποίο χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρωσό. Κυρία Τούρουνεν, σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω στα Δανέζικα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πρώτα απ' όλα για την ε, πάρα πολύ πλήρη εργασία την οποία έχετε συντάξει. Είναι δύσκολο να μπορέσει να βρει κανείς τη σωστή ισορροπία. Αυτό προσπάθησε όμως πολύ σκληρά να το πετύχει ο εισηγητής και θέλω να τον ευχαριστήσω. Επίσης και με τους σκιώδεις εισηγητές έχει προσπαθήσει να βρει συνένεση σε κάθε συγκεκριμένο σημείο. Έχουμε κάνει βέβαια τη συζήτηση σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά τώρα πρέπει να φτάσουμε και σε ένα επίπεδο λεπτομέρειες και να λύσουμε τα επιμέρους θέματα. Μπορεί αυτό να χρειαστεί πολύ χρόνο, αλλά πρέπει να προβούμε και σε αυτό το εγχείρημα. Αν δούμε λοιπόν τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικά και θετικά δικαιώματα για τους ε, καταναλωτές. Πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε οι προσόφερες των καταναλωτών τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς για να μπορούν να έχουν λογικές τιμές. Αυτό πρέπει να το εξασφαλίσουμε και να το επιτύχουμε. Υπάρχουν τώρα διαφορετικά υποδείγματα. Είναι κάτι το οποίο είναι αποφασιστικό για τους πράσινους. Εμείς θέλουμε να έχουμε μοντέλα τα οποία να λειτουργούν στην πράξη. Η κυρία Γουάλης από την Επιτροπή ε, νομικών θεμάτων ήταν πολύ συχνά στην Επιτροπή μας για τα θέματα αυτά και έπαιξε σημαντικό ρόλο. Και εγώ είμαι νομομαθής, αλλά είναι τόσο πολύπλοκα τα ζητήματα αυτά σε σχέση με το εθνικό ενοχικό δίκαιο. Κάποια πράγματα εδώ γίνονται ουσιαστικά με, αντίθετο, με αντίθετη σειρά από ότι στο εθνικό δίκαιο. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να εξασφαλίσουμε την ισορροπία. Για τα υποδείγματα λοιπόν τα οποία ακολουθούνται, νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε εκεί αυτό το οποίο μας λέει η νομική επιτροπή, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για την επιλογή των μοντέλων. Έρχομαι τώρα στο ζήτημα της εναρμόνισης. Ενδεχομένως, μπορούμε σε κάποιους τομείς να εξασφαλίσουμε απόλυτη εναρμόνιση. Αλλά ούτε και εκεί είμαι εγώ απόλυτα πεπισμένη. Ενδεχομένως να είναι δυνατό να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτή την απόλυτη εναρμόνιση. Αλλά αυτό θέλουμε, να έχουμε μια απόλυτα εναρμονισμένη ε, εσωτερική αγορά. Ξέρουμε ότι αυτό γίνεται όμως σταδιακά, ότι γίνεται με ένα ούτως είπιν εμβαλωματικό τρόπο, γιατί ξεκινάμε ως σημείο κίνηση από 27 χρόνια, από 27 κράτη-μέλη με διαφορετικά συστήματα. Χρειαζόμαστε χρόνο και υπομονή. Για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε λοιπόν μια πλήρη λύση σε νομοθετικό επίπεδο, είναι κάτι χρονοβόρο και κάτι που απαιτεί υπομονή. Αλλά η πλήρης εναρμόνιση δικαιολογείται μονάχα αν μας δώσει πραγματικά σημαντικά πλέον εμείς ως πράσινοι τα βλέπουμε τα πράγματα αυτά πάρα πολύ απτά και συγκεκριμένα. Δεν θέλουμε να τα δούμε θεωρητικά, θέλουμε να δούμε τι θα προκύψει για τον καταναλωτή. Όπως ελέγχθηκε στη συζήτηση με τον ε, ε με τον εκπρόσωπο της Βελικής Προεδρίας. Τι είναι η Ευρώπη και πώς πρέπει να την καταλάβει ο Ευρωπαίος πολίτης. Εγώ σκέφτομαι αυτά που έλεγε ο Ρομπέρ Σουμάνο, ότι πρέπει η Ευρώπη να λειτουργήσει συγκεκριμένα και θετικά για τον Ευρωπαίο πολίτη. Αυτή είναι η, αυτό είναι το ευρωπαϊκό πνεύμα, αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη λοιπόν που είναι απαραίτητη, η οποία θα πρέπει να λειτουργήσει για όλους. Αυτό θέλουμε λοιπόν να πετύχουμε εμείς ως πράσινη, μια πρακτική αντιμετώπιση. Και φυσικά πρόκειται για τα δικαιώματα που αφορούν το ενοχικό δικαίωμα, ε, Ανδρέας, και αυτά τα οποία αναφέρονται στο σημείο 8, τα οποία για μας είναι το ελάχιστο το οποίο θα πρέπει να επιτευχθεί. Δεν μας λέει η συνθήκη της Λισαβόνας ότι δεν μπορούμε να έχουμε μία μεικτή προσέγγιση μια πλήρη εναρμόνιση σε ορισμένου τομεί και μια λιγότερη εναρμόνιση σε άλλου τομεί. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε με ποιο τρόπο θα πιέσουμε για να υπάρχει το μεγαλύτερο επίπεδο εναρμόνισης. Είναι για μένα λοιπόν μια μεγάλη ε, ευκαιρία αυτό το οποίο έχουμε ενώπιόν μας. Για το άρθρο 4 επίσης. Είπαμε ότι θέλουμε να έχουμε μια οδηγία η οποία θα καλύψει όλους αυτούς τους τομείς και θα μπορέσει να δημιουργήσει προϋποθέσεις εναρμόνισης. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν με ένα στοχευμένο τρόπο. Το κατανοώ αυτό. Θα πρέπει λοιπόν για κάθε κεφάλαιο να έχουμε ένα πρώτο άρθρο όπου καθορίζονται ακριβώς οι στόχοι της εναρμόνισης. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό από την ε, οπτική γωνία των πρασίνων. Και επίσης θα πρέπει να πούμε πού είναι και τα πλεονεκτήματα της ε, συνολικής ε, και αυτό είναι σημαντικό ιδίως για το κεφάλαιο 3 και το κεφάλαιο 1 και ενδεχομένω και για ένα τμήμα του κεφαλαίου 4. Αλλά για τα υπόλοιπα τμήματα εμείς έχουμε μια κάπως επικριτική στάση και γι' αυτό βλέπουμε κάπως επιφυλακτικά με μερικές από τις προτάσεις του συναδέλφου του κυρίου Σουάμπ. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε όμως να βρούμε μια κοινή δομή. Αναφέρθηκε ο κύριος Ροσφόρ στην λεγόμενη δοκιμασία αποτελεσματικότητος. Και αυτό είναι πολύ σαφές στην πρόταση του κ. Σουβάπ. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση η οποία χάρη στο θετικό πνεύμα νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα επωφελής. Οι περισσότεροι από εμά μπορούμε να υποστηρίξουμε μια κοινή γραμμή η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε ισχυρά διαπραγματευτικά του έναντι του Συμβουλίου. Είναι λοιπόν σημαντικό εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξουμε τα δικαιώματα του Ευρωπαίου καταναλωτή. Γι' αυτό εγώ είμαι έτοιμη να συνεργαστώ προς την κατεύθυνση αυτή. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη συνεργασία που υπήρξε μέχρι αυτή τη στιγμή και φυσικά μετά από τις θερινές διακοπές θα πρέπει να περάσουμε σε λεπτομέρειες και στη διατύπωση τροπολογιών. Καλή τύχη λοιπόν σε όλους αυτά τα πλαίσια. Κύριος Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε πάρα πολύ σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή να συμφωνήσω μαζί του για τη στοχευμένη εναρμόνιση, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε τους τομείς που θα εφαρμοστεί αυτή η εναρμόνιση. Ε, σαν πολιτική ομάδα, εμείς πιστεύουμε ότι τα κεφάλαια 2 και 3 πρέπει να μείνουν ξεχωριστά και ένα μικρό σχόλιο σε ό,τι αφορά τη μεταφορά του κινδύνου. Ο καταναλωτής θα πρέπει πάντοτε σε κάθε περίπτωση να είναι ενήμερος και τον, να έχει τον πρώτο λόγο αν θα υπάρξει αλλαγή, αποζημίωση ή οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ. Thank you for your very sharp, um... Ευχαριστούμε για τις ε, εχμηρές σας παρατηρήσεις. Άλλοι ομιλητές τώρα. Στάιλερ, σας Μπίλτ. Κάποιος άλλος να λάβει το λόγο, προτού δώσω το λόγο στην Κομισιόν και φυσικά ο κύριος Σουάμπ για να κλείσει μετά. Η κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Μερικά σύντομα ερωτήματα. Στην ε, αιτιολογική σας έκθεση αναφερόσαστε σε ορισμένες μορφές εκχωρήσεων αρμοδιότητας. Μπορείτε να είστε πιο σαφείς εκεί. Και μετά για το άρθρο 26 που είναι σημαντικό στο Ηνωμένο Βασίλειο το δικαίωμα να απορρίψει κανείς μια προσφορά και το δικαίωμα διευκρίνησης. Υπάρχουν μερικά σημεία που θέλω διευκρίνηση καλύτερα για το άρθρο 13 όπου πρόκειται για το θέμα της περίοδου απόσυρσης από μια συμφωνία, αποχώρηση από μια συμφωνία και επίσης για το άρθρο 28, το οποίο περιλαμβάνει την ε, διετή νομική εγγύηση, ενώ στην ε, Σκοτία έχουμε πέντε χρόνια και στην Αγγλία έξι χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ήθελα να έχω κάποια σαφήνεια εκεί. Θα ήταν σημαντικό να δούμε τις ειδικέ ρυθμίσεις και να τις σκεφτούμε και να δούμε πού θα εξευρεθεί η ισορροπία την οποία θα θέλουμε να έχουμε. Αλλά ζητώ τη διευκρίνησή σας στα συγκεκριμένα αυτά σημεία γιατί αυτό θα έχει μεγάλη σημασία όταν πρέπει εμεί να καταθέσουμε τροπολογίε, να είμαστε σαφεί με τι πρόκειται και θέλω να σα ευχαριστήσω για το έργο σα μέχρι στιγμή. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές διαφορές ε, και στην Αγγλία και στη Σκοτία και το έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να υποστηρίξω τον εισηγητή για, αυτή την, για αυτά που είπε για την στοχευμένη και μέγιστη εναρμόνιση. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να προσέξουμε, να μην αποδυναμώσουμε ε, την ε, κοινή νομοθεσία. Ε, για το κεφάλαιο 5, αν έχουμε ένα κράτος μέλος ε, το οποίο βάλει μάλλον κάποιοι, αν οι χώρες τοποθετήσουν κάποιους κακούς ε, εμπόρους αν θέλετε στη μαύρη λίστα ή στην ε, γκρίζα λίστα κτλ πώς θα προστατεύσουμε τους καταναλωτές με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Νομίζω ότι θα επικρατήσει μια κάποια σύγχυση. Επίσης θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα αίτια της εξαίρεσης. Δηλαδή κάποια εξαίρεση σε κάποια κοινή νομοθεσία έχει ένα κόστος για τις επιχειρήσεις. Και αυτό το κόστος μετακυλίεται στους καταναλωτές. Ο καταναλωτής θέλει να έχει ανταγωνιστικές τιμές. Εάν έχουμε σαφείς και διάφανους κανόνες, τότε θα έχουμε και ανταγωνιστικέ τιμέ για τα καταναλωτή. Και αυτό θα πρέπει να εμφανιστεί στην έκθεση. Προφανώ λέω και στον κύριο Ροσφόρ ότι σε εθνικό επίπεδο θα γίνει συζήτηση για το τι χάνουμε αν θέλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτά τα οποία ενδεχόμενα να ίσχυαν σε, σε εθνικό επίπεδο. Όμω λόγω ακριβώ και τη κρίση θα πρέπει να υπερασπιστούμε την εσωτερική αγορά στα μάτια των καταναλωτών γιατί αλλιώ γιατί να βρισκόμαστε εδώ. Θα μπορούσαμε να υποκύψουμε όλοι σε έναν αναλαϊκισμό. Επίσης, αυτός ο αντίκτυπος στο εθνικό επίπεδο προστασίας καταναλωτή ε, έχουμε και την αρχική πρόταση της Κομισιόν του 2009 που νομίζω ότι είναι ένας καλός τρόπος για να προχωρήσουμε. Στο άνθρωπο 13 ο εισηγητής από τους τρεις μήνες πήγε σε έναν χρόνο, δηλαδή συνδυάζει την πρόταση της, για, την, ελάχιστη, για την κοινή αν θέλετε νομοθεσία στα υψηλότερα πρότυπα και δεν ξέρω αν δεν είμαι καλά ε, ενημερωμένη, αλλά νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος τρόπος για να προχωρήσουμε, για να ε, καταγράψουμε αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε ουσιαστικά για την προστασία των καταναλωτή και να τα προτείνουμε έτσι ώστε να είναι κοινά πρότυπα και να μην συνεχίσουμε αυτές τις εθνικές, εθνικιστικές ή λαϊκιστικές συζητήσεις για το ποιος είναι καλύτερος. Ευχαριστώ, ο κύριος Άμπατ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Ανδρέα Σβάμπ για, για την έκθεσή του και για, τα θέμ, και για τις εξηγήσεις που μας έδωσε. Ε, νομίζω ότι εξελίσσεται κάθε φορά. Ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά την προσέγγιση. Έχουμε την εντύπωση ότι προτιμάμε να έχουμε μια ε, νομική αντιμετώπιση και όχι τόσο πολιτική. Ε, Γι' αυτό ακριβώ το λόγο εμεί θεωρούμε με τους συναδέλφου Ζουβάν και Λεγκρίπο ότι αυτή η οδηγία θα βελτιώσει την κατάσταση με, αν λάβουμε υπόψη μα δύο θέματα. Το ένα είναι οι διασυνοριακέ συναλλαγέ και το δεύτερο είναι η προστασία του καταναλωτή. Θα πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση πολύ πιο ευρωπαϊκή και όχι μια εθνική προσέγγιση. Θα πρέπει να αλλάξουμε κάποια θέματα ε, Κυρίω όσον αφορά την προστασία του, βελτίωση προστασία του καταναλωτή. Και είναι απαραίτητο να έχουμε και μια πιο πραγματιστική προσέγγιση, όπω είπε και ο Ρομπέρο Φορ προηγουμένω, γιατί υπάρχουν πολλά στοιχεία στο εθνικό δίκαιο, ξέρω το γαλλικό δίκαιο καλύτερα, αλλά και σε περιπτώσει άλλων χωρών, που δεν εφαρμόζονται πλήρω αυτέ οι ρήτρε και επομένω θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι πρακτικέ απόρριε για μια τέτοια οδηγία. Εγώ νομίζω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει πέρα της προστασίας του καταναλωτές και κάποιο, κάποια δοκιμασία αντοχής στην ίδια την αγορά. Και να ξέρουμε τι ακριβώς περιλαμβάνουν αυτές οι διασφαλίσεις και ποιες είναι οι πραγματικές πολιτικές επιλογές που θα πρέπει να γίνουν από τα κράτη-μέλη για να εξασφαλιστεί αυτή η προστασία. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε τα θέματα μονάχα <clears throat> υπό την έποψη μονάχα μιας ισορροπίας, δηλαδή να βελτιώνται κάποια πράγματα ενώ άλλα επιδεινώνται. Αυτό θα οδηγήσει σε μια απόρριψη από την πλευρά των πολιτών. Είναι σημαντικό για μας λοιπόν να έχουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα για να καταδείξουμε αυτή την προσέγγιση. Με τους συναδέλφους μου Ζουβέν και Λεγκρίπ Έχουμε αντιμετωπίσει μια σειρά τέτοια, τέτοιων θεμάτων. Ξέρω ότι σήμερα τα συμβόλαια εξ αποστάσεως έχουν μια διαφοροποιημένη αντιμετώπιση από τα συμβόλαια που γίνονται πρόσωπο με πρόσωπο και αυτό οδηγεί σε προβλήματα στην ε, ανάκτηση πληρωμών μετά από την ε, κατά τη διάρκεια της περίοδου αποχώρησης. Θα ήθελα επίσης να ξέρω ποια είναι η σχέση μεταξύ του άρθρου που αναφέρει τι είναι καταχρηστική ρύθμιση και του άρθρου 32, αν θα υπάρξει περαιτέρω διευκρίνηση στην έκθεσή σας για τα θέματα αυτά και φυσικά θέλω να τονίσω ότι σημειώσαμε απόλυτα το νέο διάγραμμα που έχετε προτείνει. Υπάρχουν άλλες, άλλοι συνάδελφοι που να πάρουν το λόγο να κάνω και κάποια σχόλια, αν μου επιτρέπετε. Καταρχάς, να πω, δεν μας έχεις πει ακόμα, Ανδρέα, το χρονοδιάγραμμα επίσημα. Ίσως να το ξεκαθαρίσουμε αυτό καταρχάς. Αυτό. Μετά την τόσο πετυχημένη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών την προηγούμενη εβδομάδα, που συνέχισε την συζήτηση των θεμάτων που είχαμε θίξει στην πρώτη μας συνάντηση, ο εισηγητή πρότεινε μεγαλύτερες προθεσμίες, αν θέλετε, στο χρονοδιάγραμμά μας πρότεινε και συνάδελφος να το πάρουμε το, το κείμενο αυτό μαζί μας στις διακοπές, στην παραλία και να το συζητήσουμε και να το σκεφτούμε, να δούμε τι δικαιώματα έχουμε. Τέλος πάντων. Είναι 110 σελίδες η έκθεση αυτή, αλλά έχουμε πολύ δουλειά να κάνουμε. Ούτως ή άλλως. Υπάρχουν πολλές προτάσεις ε, για τις οποίες θα ήθελα να σας ενημερώσω και για τις οποίες συμφώνησαν οι σχεώδεις συγητές. Καταρχάς, όταν επιστρέψουμε μετά το, τις διακοπές του Αυγούστου, στις 2 Σεπτεμβρίου θα λάβει χώρα μια έκτακτη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών που θα συζητήσει τα θέματα που συζητήσαμε και τόσο στο Στρασβούργο. Και αφού... Και, ε, θα είναι στην ίδια αίθουσα που θα ε, ψηφίσουμε την έκθεση Ρουιλέ, αλλά θα είναι μια ε, και των θυρών συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. και μετά θα, υπάρχει, θα υπάρξει μια προθεσμία μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα, για την υποβολή των τροπολογιών. Στις 18 ε, Νοεμβρίου ε, θα συζητήσουμε τις τροπολογίες και στις 9 Δεκεμβρίου θα υπάρχει ε, η ψήφιση της έκθεσης στην Επιτροπή. Το ακούσατε και από τη Βελγική Προεδρία, ε, που νομίζω ότι θα συνεχίσουν τις ε, επαφές τους ε, και με τον εισηγητή και με τους σκιώδεις εισηγητές για να προχωρήσουμε, γιατί όντως υπάρχει ανάγκη να συζητηθεί το θέμα και να προχωρήσει. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, έχει δημιουργήσει πολλές διαφωνίες, αλλά πιστεύω ότι και στην Επιτροπή ε, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και θα μας μιλήσει για αυτά ο κύριος Σπρόγκ. Τώρα παίρνω το λόγο και σαν τη Επιτροπή, αλλά και σαν σκιώδη ηγητή ε, για να σας πω ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου τι συνέπειες και τα πλεονεκτήματα αυτής της πρόταση. όπως πάρα πολλοί συνάδελφοι είπαν όφελο των καταναλωτών η έκθεση αυτή, αλλά Εάν δούμε και την έκθεση αντικτύπου της Κομισιόν, και αυτό έγινε στην προηγούμενη θητεία, η έκθεση αυτή ήταν, έλεγε ότι θα έπρεπε να βελτιώσουμε το κλίμα για τις διασυνοριακές υπηρεσίες. Και αυτή είναι μια ισορροπία την οποία θέλουμε να πετύχουμε ακόμα, διότι εάν δεν υπάρχει μια σημαντική προστιθέμενη αξία της πρότασης αυτής, το κόστος εισαγωγής αυτών των προτάσεων και η περιπλοκότητα των προτάσεων αυτών και η έλλειψη ενός σαφούς πλαισίου ε, μέσα στο οποίο οι καταναλωτές να μπορέσουν να εφαρμόσουν τα, τα δικαιώματά τους, ε, δεν θα μας βοηθήσει σε τίποτα. Δεν θα οδηγήσει πουθενά. θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια εναρμόνιση, χωρίς όμως να θέσουμε τους καταναλωτές σε δυσμενέστερη θέση. Γι' αυτό ίσως θα έπρεπε να στοχεύουμε ε, σε τομείς όπου μπορεί να υπάρξει μια επιτυχημένη ισορροπία, αν θέλετε. Ε, και εδώ θα πρέπει να ζητήσουμε και τη βοήθεια της Κομισιόν. Θα πρέπει να ε, εξετάσουμε την ανάλυση που έκανε και η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ ε, και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία, να δούμε ποιοι είναι οι τομείς όπου θα μπορούσαν να βελτιωθούν αυτές οι διασυνοριακές υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη το online business και ε, να σας υπενθυμίσω ότι η έκθεση αντικτύπου και η έκθεση συνεπειών αναφέρεται στα θέματα ε, που θίγει η συνθήκη της, των Βρυξελών, η Σύμβαση των Βρυξελών. υπάρχει πρόσβαση σε κάποιες υπηρεσίες ε, από πλευρά των καταναλωτών, ανάλογα στην χώρα που ζουν. Α, όχι, δεν ήταν η σύμβαση της, των Βρυξελών, η σύμβαση της Ρώμης, αλλά τέλος πάντων τα μπέρδεψα λίγο. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι όλοι σας καταλάβατε γιατί μιλούσα. Τέλος πάντων, αυτό το οποίο προτείνω είναι να έχουμε ένα πλαίσιο με διάφορες ε, εναλλακτικέ λύσεις ε, που, μπορεί, που υπάρχουν, έτσι ώστε να κάνουμε τις σωστές επιλογές και να αποφασίσουμε πώς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το φάκελο αυτό, αλλά και την καινούρια δομή που προτείνει ο εισηγητής. Και ολοκληρώνω λέγοντας ότι θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο 6, διότι είναι πάρα είναι ξεκάθαρο, είναι σαφές, ότι αυτό το, αυτό εδώ το πακέτο για, για την προστασία του καταναλωτή είναι ένα κομμάτι ενός γενικότερου πακέτου που έχει σαν στόχο την, ε, ε, να βοηθήσει τους καταναλωτές να εφαρμόσουν τα δικαιώματά τους. Και στο άρθρο 6 υπάρχουν ε, πολλές προτάσεις για το πόσο θα αποφύγουμε ένα περαιτέρω κατακαιρματισμό. Ξέρω ότι ο κύριος Ντάλι και σαν διευθυν, Επίτροπος ε, υπεύθυνο για τα θέματα καταναλωτών θέλει να εξετάσουμε από στρατηγικής πλευράς ε, την πρόταση αυτή και ελπίζουμε ότι θα τα δούμε όλα αυτά πριν καταλήξουμε στα συγκεκριμένα συμπεράσματα και στην ε, ψηφοφορία. Αυτά, τα, αυτά ήθελα να πω και εγώ σαν πρόεδρος, αλλά και να σας πω και το χρονοδιάγραμμα, το, το οποίο νομίζω ότι ικανοποίησε όλους. Τώρα θα ήθελα να ζητήσω από τον, τον, κύριο, από τον κύριο Πρόγκ να πάρει το λόγο εξ ονόματος ε, της ε, κυρίας Ρέντινγκ, της Επιτρόπου. Και μετά θα δώσω το λόγο και στον εισηγητή για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο αλλά θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για τις προσπάθειές του, γιατί τα πράγματα γίνονται όλο και σαφέστερα και η συζήτηση δείχνει ότι οι περισσότεροι καταλαβαίνουν τις κύριες κατευθυντήρες γραμμές της συζήτησης. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Πιστεύουμε ότι το σχέδιο έκθεσης αποτελεί μια πολύ καλή βάση για συμβαστική λύση και ήδη έχει αντιμετωπίσει πολλές από τις ε, ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα που έχουν ε, αναφερθεί σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν. Παραμένουν φυσικά πολλές τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες παραμένουν αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κάποιο μεταγενέστερο στάδιο αυτές οι λεπτομέρειες. Όχι τώρα. Το βασικό είναι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για μια γενική προσέγγιση η Κομισιόν μπορεί να υποστηρίξει τις προτάσεις του εισηγητή για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να προχωρήσει σε εναρμόνιση των ορισμών και την ε, συγχώρευση του κεφαλαίου 2 και 3 σε ένα κεφάλαιο για τις ανάγκες πληροφόρησης και τις προϋποθέσεις αποχώρησης από μια σύμβαση και επίσης αυτά που θέλει να διατηρήσει για τις ε, συμβάσεις που γίνονται on-premises όπως λέγεται, όπου τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν τις ισχύουσες ρήτρε. Και για το κεφάλαιο 5 να εξασφαλίσει για τα κράτη-μέλη ελευθερία σε σχέση με τις συμβάσεις οι οποίες θεωρούνται μη δίκαιες ή καταχρηστικές και επίσης για την πρόθεση της εναρμόνισης στο κεφάλαιο 4. Όλα αυτά λοιπόν είναι αποδεκτά από την πλευρά της Κομισιόν θα πρέπει φυσικά όλα αυτά να αποτελέσουν και αντικείμενο διαπραγμάτευση μεταξύ των εμπλεκομένων εταίρων στην διαδικασία νομοθετικής συναπόφασης. Τα επιμέρους τώρα ερωτήματα δεν είναι πολύ εύκολα. Καταρχήν για το άρθρο 4. Για το άρθρο 4 ως έχει και εδώ θα πρέπει να λάβετε υπόψη την πρόταση της Κομισιόν, που ζήτησε πλήρη εναρμόνιση η Κομισιόν. Το άρθρο 4 είχε απόλυτη λογική μέσα στο πλαίσιο αυτό. Από την πλευρά του εισηγητής ο κ. Σουάπ προτείνει μια στοχευμένη εναρμόνιση. Το δικό του άρθρο 4 λοιπόν είναι και αυτό λογικό γιατί δεν μπορούν όλα να καλυφθούν από πλήρη εναρμόνιση κατά την άποψή του. Αν προχωρήσουμε όμως ένα βήμα περισσότερο, μπαίνουμε σε ένα προβληματικό χώρο, αν θέλετε να το θέσω έτσι. Γιατί? Γιατί υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της πλήρους εναρμόνσης και της εξελαχίστων εναρμόνσης. Η μίνιμουμ εναρμόνιση είναι ουσιαστικά δημιουργία προτύπων, το οποίο σημαίνει ότι φυσιολογικά καταλήγει κανείς σε ένα επίπεδο που είναι πολύ κοντά σε αυτό το οποίο ισχύει στα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη-μέλη. Γιατί άμα ζητηθεί κάτι περισσότερο θα αρχίσουν να διαμαρτύρονται. Αυτό γίνεται συνέχεια στο Συμβούλιο. Η πλήρης εναρμόνιση σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσουμε στο επίπεδο του πιο προωθημένου κράτους. Γιατί δεν θέλει κανείς να χάσει τα δικαιώματα τα οποία έχουν αποκτή, αποκτηθεί. Δεν μπορείτε όμως να αναμίξετε τα δύο ως εάν ή το μια ανάμιξη αμνών με ερυφιάκια. Αν έχετε πλήρη εναρμόνιση μπορείτε να αποχωρήσετε περισσότερο προς υψηλότερα πρότυπα και δημιουργείτε τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς. Η εσωτερική αγορά ευνοεί τη χρήση από τους εμπορευόμενους των δυνατοτήτων που δίνει η πλήρης αγορά. Ξέρουμε όμως ότι πολλές χώρες δεν μπορούν να είναι προμηθευτές μέσω του διαδικτύου, διότι υπάρχουν διαφορές σε νομικό επίπεδο, σε νομοθετικό επίπεδο, στις ρυθμίσεις. Όταν έχουμε λοιπόν ελάχιστη εναρμόνιση, αυτό δεν δημιουργεί μια κατάσταση θετικού αθροίσματος. Δεν ενδιαφέρει τους προμηθευτέ να χρησιμοποιήσουν όλη την αγορά. Με ελάχιστη εναρμόνιση παραμένουμε σε ένα χαμηλότερο επίπεδο και δεν αποκομίσουμε το πλήρες όφελος από την διάσταση της εσωτερικής αγοράς. Η κυρία Μπίλτ μας ρώτησε για αυτό το θέμα. Μπορώ να σας παραπέμψω στην παλιά μας έκθεση αντικτύπου, μελέτη αντικτύπου και εκεί φαίνεται τι θα προκύψει αν αφήσουμε μερικά ζητήματα έξω από την εναρμόνιση. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε μια νέα μελέτη αντικτύπου, ίσως όμως μπορούμε να σας δώσουμε κάποια στοιχεία επί τη βάση της προηγούμενης μελέτης αντικτύπου πριν από τη διατύπωση της οδηγίας. Για την Κομισιόν λοιπόν θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τροποποιήσουμε το σύστημα του αρθρού 4. Απόλυτα. Γιατί με τον τρόπο αυτό η Κομισιόν θα έχανε τα μάλα και δεν θα συνέβαλε ούτως ή άλλως πια το άρθρο 4 στην διαμόρφωση της εσωτερικής αγοράς. Αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο να το αποδεχτούμε. Υπήρξαν κάποια ερωτήματα σε σχέση με το ποια είναι τα ωφέλη τα οποία θα αποκομιστούν σε περίπτωση πλήρους εναρμόνισης. Υπήρχε ένα πολύ καλό παράδειγμα στην αρχή για τη χάρτα δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών. Φανταστείτε ότι ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα μπαίνετε σε ένα αεροπλάνο στις Βρυξέλλες και ξέρετε ποια είναι τα δικαιώματά σας. Αλλά αν έρχεστε από μια άλλη χώρα, ξέρετε τι γίνεται στη δική σας χώρα, αλλά δεν ξέρετε αν στο Βέλιο ισχύουν τα ίδια αυτά δικαιώματα όταν φτάσετε στο Ζάβετε. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι ένας καταναλωτής σε ένα κράτος μέλος γνωρίζει ποια είναι τα δικαιώματά του, μόλις φύγει όμως από τα σύνορα, αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει ποια είναι τα δικαιώματά του. Μόνο αν είναι εναρμονισμένα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ξέρει ποια είναι τα δικαιώματά του. Και φυσικά αυτό είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα. Το άλλο είναι η, η προμήθεια αγαθών. Ξέρει η Κομισιόν ότι αν υπάρξει μεγαλύτερη αναρμόνιση θα τονωθεί η προσφορά αγαθών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα είναι τελικά θετικό για τους καταναλωτές το να μπορούν να παίρνουν αγαθά τα οποία δεν μπορούν να βρουν κάπου αλλού. Επομένως το άρθρο 4 είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να δείτε κανείς όλες τις δυνατότητες αλλά το να αφήσουμε την πλήρη αναρμόνιση εκτός του άρθρου 4 θα δημιουργήσει μια κατάσταση που να μην είναι ιδιαίτερα πρόσφορη για τους ε, προμηθευτές. Και αυτό θα είναι κρίμα. Για τα νομικά τώρα ζητήματα που εγέρθηκαν πρέπει να δούμε το τελικό κείμενο για να μπορέσουμε να τα εκτιμήσουμε αυτά τα νομικά σημεία. Είναι γεγονός ότι η νομική βάση μιλάει για την προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών. Αυτό λέει το αντίστοιχο άρθρο. Αν δεν προκύψει κάποια προσέγγιση, τότε είναι δύσκολο το θέμα της νομικής βάσης. Αλλά δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε το κατά πόσον θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει προσέγγιση αυτή τη στιγμή. Εγώ θα σας έλεγα ότι δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ξέρουμε βέβαια ότι η νομική βάση Ήτανε καταρχήν επαρκής για αυτή την οδηγία. Αν αλλάξει όμως εκβάθρον αυτή η οδηγία, είναι πιθανόν ότι δεν θα επαρκεί. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ότι απάντησα τα ερωτήματα. Και φυσικά η Κομισιόν είναι πάντα έτοιμη να βοηθήσει, να σας βοηθήσει, σε ό,τι αφορά όμως τα αριθμητικά στοιχεία Έχουμε μονάχα αυτά από την προηγούμενη μελέτη αντικτύπου. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό σαν σημείο εκκίνησης και είναι αδύνατον μέσα στον απαραίτητο χρόνο, στον ελάχιστο χρόνο που είναι ενώπιόν μας να έχουμε πλήρη στοιχεία. Μόνο μερικά επιμέρους στοιχεία έχουμε και την παλιά έκθεση αντικτύπου. Okay, well, um, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ακούσαμε διάφορα πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν και τον Ανδρέα Σουάμπα για την ε, έκθεση των συνεπειών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, τις συνέπειες και τον αντίκτυπο κάθε επιμέρους μέτρου και ίσως να ε, μην ζητήσουμε νέα ανάλυση, αλλά απλώς μια ανάλυση, πιο λεπτομερή ανάλυση των, των μέτρων εναρμόνησης. Εάν και εσείς και η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ μπορείτε να μας βοηθήσετε, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Επίσης, μας είπε και ο υπουργό νωρίτερα για το πόσο η Βελγική Προεδρία θέλει να συνεργαστεί μαζί μας και ο κύριος Έντελχοφ από τη Βελγική Προεδρία είναι ακόμα μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα συμμετέχει στις συζητήσεις. Ανδρέα Βάμπ, θέλεις να κάνεις κάποιες τελικές παρατηρήσεις σου πριν ε, πάμε όλοι διακοπές. Τόσο ενθουσιασμένοι με τις λύσεις που θα βρούμε για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Έχω σημειώσει έξι συνολικά θέματα ώστε να μην μακρηγορήσω. Πρώτα για το χρονοδιάγραμμα. Όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, συμφωνήσαμε διότι οι συνάδελφοί μου έχουν θεωρήσει την πρόταση ακόμα άγνωστη για αυτούς και ε, τόσο πλούσια σε λεπτομέρεια ώστε χρειάζεται ακόμα μελέτη. Πάντως όλοι οι οδησηγητές έχουν συμφωνήσει στον κοινό στόχο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, δηλαδή εντός Βελικής Προεδρίας, να καταλήξουμε σε μια πολιτική συμφωνία πλαίσιο. Άρα η αναβολή του χρονοδιαγράμματος δεν σημαίνει ότι μειώνονται οι φιλοδοξίες μας σε ό,τι αφορά ε, την ολοκλήρωση προσπάθειας μέχρι τέλους του έτους. Θα ήθελα παρακαλώ αυτό το σχόλιο μου να εγγραφεί στο πρακτικό της σημερινής συνεδριάσεως διότι απηχεί την κοινή άποψη όλων των συνεισηγητών. Τώρα για την νομική βάση. Κυρία Τούν, εγώ απλώς επεσήμανα ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και η πρόταση δική μου βασίζονται στο άρθρο 114 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης και ότι προ λίγων ετών το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην απόφασή του για την οδηγία περί καπνού είχε πει ότι μια ελάχιστη εναρμόνιση και τότε ήταν το δίκαιο της διαφήμισης για τον καπνό μπορεί να ισχύσει εάν δεν υπάρχει άλλη προσέγγιση των νομοθετικών συστημάτων. Υπάρχουν και άλλες νομικές βάσεις. Δεν είναι πρόβλημα αυτό για μένα αλλά δεν μπορεί κανείς να επιλέξει εντός των πλαισιών του άρθρου 114. Θα πρέπει να ληφθεί ως βάση το άρθρο 114, το άρθρο για την ε, προστασία των καταναλωτών. Αλλά βέβαια με την συνδρομή της νομικής υπηρεσίας θα βρούμε τη λύση. Τώρα, την μελέτη ανακεφάλαιο. Εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και εξετάσουμε το ενοποιημένο έγγραφο, θα δούμε στο άρθρο 4 ποιο, ποια θα πρέπει να είναι η βασική αρχή. Και μετά λέει παράγραφος 1α, 1β, 1γ και εκεί εξηγείται ποια θα είναι η ρύθμιση ανακεφάλαιο. Τώρα μπορούμε βέβαια να διαφωνήσουμε και για το κάθε κείμενο της κάθε υποπαραγράφου. Αλλά εάν θέλουμε να πούμε αν θέλουμε να πούμε το 4 1 α να μπει στο άρθρο 2, το 4 1 β στο ε, κεφάλαιο 4 και το 4 1 γ στο κεφάλαιο 5, νομοτεχνικά νομίζω αυτό έχει απλώς καλοπιστικό χαρακτήρα και κανένα ουσιώδη χαρακτήρα. Δεν κατανοώ λοιπόν πολύ καλά την πρόταση. Επίσης τα αυτά που λέει ο κύριος Οσφόρ για το άρθρο 4. Μπορώ να συμφωνήσω σε ό,τι αφορά την διαδικασία. Και βέβαια η πλήρη συναρμόνιση αποτελεί μια διαδικασία και θα πρέπει και εμείς και οι οργανώσεις καταναλωτών και οι χώρες μέλη να έχουμε τον αναγκαίο χρόνο ώστε να διαμορφώσουμε τη διαδικασία αυτή με τον σωστό τρόπο. Το ερώτημα είναι αν θέλουμε να βάλουμε ένα στόχο, το οποίο, ο οποίος στόχος δεν είναι καθ' αυτόν καλός ή κακός, αλλά καθιστά απαραίτητη μια αλλαγή του status quo μόνο εάν θελήσουμε να καταλήξουμε σε μια εναρμόνιση. Επομένως το κεφάλαιο 4 δεν είναι καλό ή κακό. Λέει ότι ανεξαρτήτως των εθνικών νομοθετικών διαταξών, οι χώρες μέρη δεν έχουν δυνατότητα αλλαγή των ε, διαταξιών στον χώρο της εναρμόνισης. Δεν λέει τίποτε άλλο από αυτό. Ούτε αποτελεί μομφή σε βάρος των ε, χωρών μελών που έχουν υιοθετήσει διαφορετικές ε, ρυθμίσεις λόγω των διαφορετικών παραδοσιών τους. Ούτε άλλωστε μπορούμε να καταργήσουμε όλες αυτές τις διαφορές με την οδηγία. Και έχουμε και σε αυτή την δοκιμασία, το τεστ conformité που είπε ο κ. Ροσφόρ. Η στο αγγλικό κείμενο θα το βρείτε αυτό, λέει ότι οι χώρες μέλη μπορούν να προβλέψουν εθνικές διατάξεις κλπ. Και λέει μετά τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι ουσιώδη για να προστατεύουν τα δικαιώματα των καταναλωτών και θα πρέπει να είναι αναλογικά και αποτελεσματικά. Δεν βλέπω εδώ με ποιον τρόπο καταστρέφονται εδώ τα δικαιώματα των χωρών μελών. Και βρίσκω επίσης ότι η διατύπωση είναι σωστή. Νομίζω ότι στο άρθρο 46α γράφουμε όντως absolute necessary και αυτό νομίζω ότι είναι μάλλον μεταφραστικό σφάλμα. Εγώ νομίζω πάντως ότι μπορώ να το συζητήσουμε αυτό. Πάντως για το 26.5β νομίζω ότι η ρύθμιση είναι σωστή. και για τη σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηριού ε, σε 65 που λέει ότι η εναρμόνιση, η ελάχιστη εναρμόνιση επιτρέπει κάποια περιθώρια ελιγμών στις χώρες μέλη. Αλλά παρόλα αυτά οφείλουν να σέβονται την ενιαία αγορά και τα μέτρα που λαμβάνουν πρέπει να είναι, όπω είπα, αναλογικά και αποτελεσματικά. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να αναφερθεί εδώ η απόφαση του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τέλος, όπως είπε και ο Ροσφόρ, η οδηγία αυτή αλλάζει πολλά σωστό αυτό και όπως είδατε και από την επισκόπηση που έχω διανύμει. Πρόκειται για συγκριτικό πίνακα που βασίζεται σε μια σύγκριση που έχει κάνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει περιλάβει αρχικά στην αρχική της πρόταση. Εγώ έκανα τη σχετική προσαρμογή του πίνακα αυτού. Κατά τη γνώμη μου, η δική μου πρόταση αλλάζει κάπως λιγότερα από αυτά που αλλάζει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό νομίζω απηχεί και τις απόψεις των συναδέλφων μου. Και γι' αυτό και το θέμα με τη μελέτη αντικτύπου μπορεί να λυθεί με τον τρόπο αυτό. Εγώ νομίζω ότι με την οδηγία αυτή κάνουμε ένα πρώτο βήμα, πότε θα έρθει το δεύτερο βήμα αυτό δεν είναι γνωστό. Πάντως τα πλεονεκτήματα του τελευταίου βήματος θα είναι αυτά τα οποία περιλαμβάνονται και στη μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να πούμε ότι ναι μεν κάνουμε κάπως λιγότερα τώρα, παραμένουμε όμως πάνω στην οδό που έχει ήδη προδιαγράψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πάντως ε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι για τις προτάσεις, για την υποστήριξή σας και εγώ αναμένω με ανυπομονησία να ανταμωθούμε ξανά μετά από τις θερινές διακοπές. Υπενθυμίζω, εγώ θα περιλάβω και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την οδηγία περί καπνού και την ΣΕ 65-2009 και ελπίζω ξεκούραστη, μετά από τι ταινίε διακοπέ να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να βρούμε μια λύση υπό Βελγική Προεδρία. thank you very much indeed. Um, Ευχαριστούμε πολύ, Άντριο Σφαμπ. Σε ευχαριστώ για τόσο δύσκολο αυτό έργο και για το γεγονό ότι έχει διασαφηνίσει όλα αυτά τα θέματα. Κυρία Τουρίνα, θέλετε να πείτε κάτι. Να ξανάρθω. Γιατί είπατε ότι είχατε προβλήματα να καταλάβετε τι εννοούσε για το άρθρο 4. Δεν είναι τεχνικό σημείο για το πού θα βάλουμε το άρθρο 4. Αυτό είναι το λιγότερο πρόβλημα. Είναι το θέμα του ποια είναι η βάση αυτής της οδηγίας. Το συζητήσαμε επίσης και στην συνάντηση με τους κοιόδης συγητές, ότι θα υπήρχαν διάφορες εκδοχές, διάφορα υποδείγματα και θα το φέρατε αυτό στην επόμενη σας ε, στην επόμενη μας συζήτηση. δεν ήταν σωστό αυτό που είπατε νομίζω απόλυτα. Εντάξει, εντάξει, ναι, ναι, αυτό είχαμε συμφωνήσει, λέει ο κύριος Χάρμπορ. Και το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να βρούμε και κάποια λύση για τις δομικές αλλαγές που θέλετε να επιφέρετε στο κείμενο, τώρα που έχουμε μια σαφή επισκόψη της κατάστασης. Προφανώς δεν θα δεχτούν όλοι τις ιδέες σας, αλλά ο στόχος μας μετά τις διακοπές είναι να μπορέσουμε να δούμε ποια ακριβώς στρατηγική θα ακολουθήσουμε και μετά θα μπορέσουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις λεπτομέρειες. Και φαντάζομαι ότι και ο Επίτροπος θα είναι, ή Επίτροπος θα είναι παρόν, ή ο Επίτροπος θα είναι παρόν στη συνάντησή σας, ιδίως αν έχουμε κάποια στοιχεία, αν έχει κομισιόν κάποια στοιχεία, Προφανώ θα γίνει κάτι τέτοιο, λέει ο κύριο ε, Σουάμπ. Η δυσκολία για το άρθρο 4 είναι ότι θέλουμε να πετύχουμε πολλαπλού στόχου με αυτό το άρθρο. Θέλουμε να δώσουμε πολιτικά μηνύματα ότι η απόλυτη εναρμόνιση πρέπει να γίνει να είναι ο βασικός στόχος, αλλά ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές συνέπειες σε περίπτωση εναρμόνισης κατ ελάχιστο. Έχουμε λοιπόν μία σειρά από διαφορετικές έννοιες και εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να το δούμε αξιολογικά μονάχα τις διαφορές αυτές των απόψεών μας. Εγώ, όπως ελέγχθη, τόνισα ότι δεν πρέπει σαν αρχή να γίνει δεκτή η εκ των ελαχίστων εναρμόνιση. Εάν υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις, εγώ θα είμαι πρόθυμος να προχωρήσω σε μία συμφωνία. Ξέρω ότι δεν μπορώ εξ αρχής να κάνω μια πρόταση η οποία θα γίνει αποδεκτή από όλους και γι' αυτό αναφέρθηκα στη χρήση του άρθρου 4 προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ, λέω πρόεδρος. Ας κλείσουμε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστώ πολύ, Άντερ, Ανδρέα. Και στις 2 Σεπτεμβρίου θα επανέλθουμε. Ένα ακόμα θέμα έχουμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μην εξαφανιστείτε. Ερχόμαστε στον προϋπολογισμό προπαρασκευαστική εργασία για μια ψηφοφορία που θα πρέπει να γίνει και αυτή στις 2 Σεπτεμβρίου. Χαίρομαι που η κυρία Ρίλε είναι εδώ για να μας παρουσιάσει το θέμα αυτό. Ο κύριος Βαντερκάμπ είναι εδώ. Ο κύριος Βαντερκάμπ Πανταχούπαρο είναι εδώ. Κάποιοι άλλοι δεν είναι παρόντες, δεν ξέρω ποιος θα εκπροσωπήσει σοσιαλιστές στη συζήτηση. Κυρία Στάιλερ, ο κύριος Μπουζόιλ είναι εδώ, ο κύριος Μπίτεν δεν είναι εδώ. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης δεν είναι πια εδώ. Κυρία Ρούλα έχετε το λόγο λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Θα το κάνουμε σύντομα και συνοπτικά. Θέλω να ευχαριστήσω, θέλω μάλλον θέλω να πληροφορήσω όλου του συναδέλφου για κάτι πάρα πολύ θετικά. Πήραμε την προηγούμενη εβδομάδα την απάντηση τη Κομισιόν για την πρότασή μα σε σχέση με τα πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικέ δράσει. Αυτό το οποίο είναι θετικό είναι ότι η προπαρασκευαστική δράση για την παρακολούθηση μέτρων στον τομέα της πολιτικής καταναλωτών και για μας συνάπτεται αυτό με το λεγόμενο scoreboard. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει δεχτεί η Κομισιόν και έχει υποστηρίξει την πρότασή μας. Έχει επίσης υποστηρίξει την πρότασή μας να υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για το φόρουμ της εσωτερικής αγοράς. Και αναφέρεται στο ότι ορισμένα από αυτά τα θέματα που άπτονται των σχέσεων με την Κομισιόν έχουν ήδη καλυφθεί και επομένως δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμα το να προχωρήσουμε σε αυτό το πιλωτικό σχέδιο. Μπορούμε να βρούμε ίσως κάποια συμβιβαστική λύση και εγώ θα θεωρούσα ότι η λύση θα ήταν να δώσουμε μια μεγαλύτερη έμφαση στο φόρουμ της εσωτερικής αγοράς. Η Κομισιόν έχει αναφέρει τη σημασία της εκδηλώσεως της 9ης Νοεμβρίου και τόνισε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα φόρουμ στο οποίο να είναι σε πιο <clears throat> μεγάλο βαθμό εμπεπλεγμένοι οι καταναλωτές και οι πολίτες και επομένως νομίζω ότι το φόρουμ αυτό για την, ενωμένη, την ενιαία αγορά μπορεί να έχει ένα επιτυχή ρόλο και μπορούμε με αυτή τη μορφή να το παρουσιάσουμε ως πιλωτικό πρόγραμμα. Και φυσικά το φόρμα αυτό θα δώσει μια προσθέμενη αξία για τους καταναλωτές και για τους, πολ... και για τους πολίτες. Θα πρέπει μέσα στα πλαίσια της δράσης μας, επομένως χρηματοδοτώντας αυτό το πρόγραμμα, να καταδείξουμε ότι εμείς υποστηρίζουμε τους καταναλωτές και τους πολίτες. Επίση, θα έχουμε ήδη μέσα σε αυτή τη βδομάδα, ελπίζω, την απάντηση του Συμβουλίου και θα ξέρουμε κατά πόσο το Συμβούλιο θα απορρίψει τις προτάσεις της Κομισιόν. Αυτό το οποίο μπορεί να είναι προβληματικό είναι ότι μπορεί να περικόψει δραστικά τις ε, πιστώσεις για τα προγράμματα αυτά. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία έχουν μακρά χρονική διάρκεια και χρειάζονται ήδη μια χρηματοδότηση για αυτό το διάστημα και αν υπάρξουν σημαντικές περικοπές στις πιστώσεις πληρωμών θα είναι προβληματική συνέχιση αυτών των ε, προγραμμάτων. Γι' αυτό πρέπει να συνεργαστούμε με την Επιτροπή Προπολογισμών, να εξασφαλίσουμε ότι θα απορριφθούν οι θέσει του Συμβουλίου και θα επανέλθουν οι προτάσει τη Κομισιόν, αλλά είναι απαραίτητο για να κάνουμε κάτι τέτοιο να έχουμε και καλέ προτάσει και να έχουμε και την σύμπραξη των πολιτών μα. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να γίνουν μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο όπου έχουμε τα προβλήματα των υπερχρεωμένων κρατών μας, γενικά του προβλήματος της οικονομικής κρίσης. Είναι λοιπόν απαραίτητο να τονίσουμε ότι οι προτάσεις μας έχουν σημασία για την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές, για την εποπτεία της αγοράς, ότι είναι προτάσεις από τις οποίες θα μπορέσουν να υποφελθούν κατευθείαν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπατε όλα αυτά με τέτοια σαφήνεια. Ο κύριος Κάμπ αναφέρθηκε και στις επιχειρήσεις που νομίζω ότι και αυτό αντικατοπτρίζεται εδώ. Και όπως είπατε βέβαια και εσείς θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν εγκαίρως. Ας ακούσουμε από τους σκιώδεις εισηγητές και μετά να δούμε και το χρονοδιάγραμμα. Ο κύριος Κάμπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ρούλε, την συνάδελφό μας, για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Ε, το πήραμε λίγο με κάποια καθυστέρηση, οφείλω να πω, αλλά καλύτερα τώρα παρά ποτέ. Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με αυτά τα οποία προτείνει η κυρία Ρούλε. Αυτό όμως ε, το οποίο δεν καταλαβαίνω πολύ καλά είναι πώς θα υποβάλουμε τις παρατηρήσεις μας στο Συμβούλιο. Καθαρά τεχνικής φύσης ε, η απορία μου. Και τελευταία παρατήρηση το χρονοδιάγραμμα. Πρέπει να υποβάλουμε τις τροπολογίες μέχρι τις 12 Αυγούστου. Όμως τότε όλοι θα λείπουν για διακοπές. Τι θα κάνουμε τότε. Ευχαριστώ. Um, Κύριε Καπ, δεν έχουμε κάποια κάποιο συγκεκριμένο προ χρονοδιάγραμμα. Το, αυτό που μας ε, πιέζει, αν θέλετε, και μας δεσμεύει είναι όλη η διαδικασία του προπολογισμού. Θα πρέπει να επανέλθουμε ε, στην, στην, μας, θα μας ξεκαθαρίσει η κυρία Ρούλε, αλλά στις 2 Σεπτεμβρίου θα γίνει μια συνάντηση για να ψηφίσουμε. Ε, επομένως θα πρέπει να έχουμε ξεκαθαρίσει όλα μέχρι τότε. Κυρία Ρούλε. Είναι σαφές ότι ο χρόνο είναι περιορισμένο και ότι κανένα να καθίσει στι νέε διακοπέ να διαβάζει τον προπολογισμό. Αλλά στι 30 Αυγούστου να κάνουμε μια συνάντηση των σκιωδών και να εξετάσουμε τι τροπολογίε. Δεν νομίζω να υπάρχουν μεγάλε συγκρούσει μεταξύ των πολιτικών ομάδων, ούτε νομίζω ότι χρειάζεται να μεταφραστούν όλε τι τροπολογίε σε όλε τι γλώσσε. Αν συμφωνήσουμε όλοι σε μια γλώσσα εργασία στα αγγλικά και μπορούμε να συνεννοηθούμε στα αγγλικά σε αυτή τη συνάντηση των σκιωδών, ε, μπορούμε νομίζω τότε να τα καταφέρουμε χωρίς να παραζοριστούμε στις διακοπές. Εγώ πολύ ευχαριστώ πάντως να συμβάλλω και εάν εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη αργότερα μπορούμε να δούμε και τις προφορικές τροπολογίες. Είμαι διατεθειμένη για να προβώ σε συμβιβασμούς. Τώρα για το Συμβούλιο. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Ξεκινήσαμε εκ του μηδενό. Δεν είχαμε το σχέδιο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά ήρθε το σχέδιο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τώρα σιγά σιγά αρχίζει και διαμορφώνεται η απάντηση του Συμβουλίου. Πρόκειται για μια καινούργια διαδικασία. Από τη θέση σε ισχύ της διαδικασίας Λισαβόνα, το Κοινοβούλιο πάρει νέα καθήκοντα. Έχει περισσότερο λόγο και στου τομεί αυτούς, συμμετέχει δηλαδή στη νομοθετική διαδικασία και αυτό βεβαίω μα αναγκάζει να εργαζόμαστε υπό νέου όρου, του οποίου δεν, δεν έχουμε συνηθίσει και είναι επομένω ένα είδο δοκιμασία αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα τον αριθμό, την απάντησή μα στο Συμβούλιο, ε, αυτά θα δούμε στην ψηφοφορία τη Δευτέρα Σεπτεμβρίου και θα έχουμε και τα απαραίτητα νούμερα τότε για την Επιτροπή Προπολογισμών. Αυτά βέβαια θα τα κάνουμε όταν θα έχουμε πρώτα τα νούμερα του Συμβουλίου. Ναι, Ούτω ή άλλω αυτά τα στοιχεία τα αριθμητικά που αναφέρατε. Τα είχαμε από ό,τι μου λέει η άλλω την προηγούμενη Παρασκευή. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τόσο εφάνταστη λύση που αναφερατε τα ειχαμε απο οτι μου λεει η γραμματεια διαθεσιμα την προηγουμενη παρασκευη αλλα σα ευχαριστω παρα πολυ για αυτη την τοσο εφανταστη λυση που δωσετε για τι τροπολογίε. Η κυρία Στάιλερ. Ο εισηγητή μα. και ο κ. Βαντερκάμπ νομίζω ότι με βρίσκουν σύμφωνοι σε μεγάλο βαθμό. Υποστηρίζουμε το σημείο 2 για την ε, πρωτοβουλία αυτή για την πρωτυποποίηση. Στο Στο σημείο 3 υπάρχουν αυτά τα οποία πολλές φορές τα ξεχνάμε. Οι διαδικασίες επιλύσεως προβλημάτων, όπως το Solvit. Εμείς υποστηρίζουμε ιδιαίτερα το Solvit ως ε, διαδικασία επίλυσης διαφορών. Και νομίζω, Χάιτι, ότι με τη διατύπωσή σου το έχεις καταφέρει να τονίσεις ότι είναι απαραίτητο το Solvit να έχει τους πόρους που χρειάζεται για να κάνει σωστά τη δουλειά του στο σημείο 4 επίση για το φόρουμ της εσωτερικής αγοράς θέλω να το υποστηρίξω είναι απαραίτητο να το υπογραμμίσεις και στο σημείο 6 ο αγώνας κατά του λαθρεμπορίου και της απάτης είναι τόσο σημαντικός για το έργο μας και πολύ ορθά και στο σημείο 8 τονίζω ότι πρέπει να συνεχίσουν οι μελέτες και οι έρευνες σε σχέση με την επισκόπηση και την εποπτεία της εσωτερικής αγοράς. Οπότε μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού νομίζω ότι έχει στήξει τα κέρια σημεία, αυτά που είναι σημαντικά και αυτά τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και γι' αυτό προσβλέπω στην ψηφοφορία της Δευτέρα Σεπτεμβρίου και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και ως Μπουζόλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά ελέγχθησαν ήδη. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος λοιπόν. Χαιρετίζω καταρχήν όλα τα σχόλια της κυρίας Ρούλας. στην, ε, στην έκθεσή τη, στην γνωμοδότησή της μάλλον και συμφωνώ απόλυτα και πιστεύω πρέπει να συνεχίσουμε με το εγχείρημά μας για το φόρουμ της εσωτερικής αγοράς. Πρέπει να το προωθήσουμε. Χαιρόμαστε που η Κόμισιόν ήταν πολύ θετική γι' αυτό. Είχαμε μια προπαρασκευαστική συνάντηση και η στάση της Κομισιόν ήταν πολύ ανοιχτή. Ίσως δεν θα ήταν λάθος να έχουμε και το δεύτερο πιλωτικό πρόγραμμα για τις αιτίε έλλειψης ικανοποίησης των καταναλωτών, το οποίο το συνδέσουμε με το φόρουμ. Λυπάμαι που εφέτος δεν έχουμε μια χωριστή γραμμή για το Solvit. Εγώ υπήρξα εισηγητής του Solvit και το Solvit είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό δίκτυο το οποίο βοηθάει τους επιχειρηματίες και τους πολίτες να γλιτώνουν λεφτά τα οποία θα ξόδευαν αν καταφεύγαν στα δικαστήρια. Δυστυχώ, πέρσι δεν καταφέραμε να έχουμε μια χωριστή γραμμή του προπολογισμού για το Solvit. Εγώ θα καταθέσω μια τροπολογία που ελπίζω θα υποστηριχθεί για να έχουμε φέτος μια χωριστή γραμμή του προπολογισμού. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σφιχτό το χρονοδιάγραμμα. Δεν θα έχουμε πολύ χρόνο με τον Σεπτέμβριο, αλλά ελπίζω ότι στο τέλος Αυγούστου στη συνάντησή μας θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια γενική συμφωνία και συνένεση και αν έχουμε μια ισχυρή συνένεση αυτό θα μπορέσει να είναι μια στεναρή στάση και γνώμη της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και ο Πρόεδρος. Κάποιες σημειώσεις από μένα μονάχα ως Πρόεδρος και ως εκπρόσωπος της ομάδας μου. Θέλω να πω ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ ισορροπημένη έκθεση από την πλευρά της κυρίας ρούρε. Λαμβάνοντας υπόψη τώρα τα σχετικά μικρά <clears throat> ποσά, μικρά κονδύλια τα οποία, διαχεί, τα οποία είναι στην αρμοδιότητα της Επιτροπής μας, πρέπει να εστιάσουμε σε, σε ενέργειες οι οποίες θα ευνοήσουν την πραγματική οικονομία. Όπως λέτε και στο άρθρο 3, θέλουμε να δώσουμε πλεονεκτήματα για την ε, ενιαία αγορά, εσωτερική αγορά εν γέννη. Γιατί είναι σε μια, όλα αυτά σε ένα πλαίσιο περικοπής των προϋπολογισμών, ενώ είναι απαραίτητο να βελτιώσουμε την εσωτερική αγορά, δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης και να δώσουμε έμφαση στο ότι η συνολική αγορά μπορεί να ενισχύεται ακόμα και αν οι τοπικές αγορές δεν προχωρούν. Για το Solvit το έχουμε υποστηρίξει πάντα στο παρελθόν και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχει την κατάλληλη χρηματοδότηση και στο μέλλον. Επομένως θα έχετε την υποστήριξή μας και για αυτό το σημείο. Χάιντι, θέλεις να πεις κάτι για να κλείσεις ή απλώς να επιβεβαιώσουμε το χρονοδιάγραμμα και τις ε, διαδικασίες που θα χρησιμοποιήσουμε και ίσως οι σκιώδεις μπορούν να παρέμουν σε άλλα θέματα. Πολύ σύντομα. Ε, θα συμφωνήσω αν κάνετε μια τροπολογία. Χωρίς πρόβλημα. Τις 30 νομίζω του μηνός θα δούμε, το Αυγούστου δηλαδή, και ατενίζω πάντως με αυτοπεποίθηση τη ε, συνάντηση της Δευτέρα Σεπτεμβρίου. Νομίζω θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Είτε με μεγάλη πλειοψηφία είτε με ομοφωνία. Right. So, um, shadows will meet on the 30th 30 Αυγούστου θα συναντηθούν οι σκιώδεις για να διευκρινίσουν τα θέματα των τροπολογιών. Αν ε, θέλετε να καθίσετε τροπολογίες μέχρι τότε, θα έχετε τη, τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Δεν ξέρω τώρα αν η Κομισιόν έχει εμπειρογνώμονες του προϋπολογισμού, επομένως η Κομισιόν δεν νομίζω ότι θα λάβει το λόγο. Θέλω να σας ευχαριστήσω, Χάιντι, πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε σε αυτό το σημείο με μεγάλη επιτυχία και προσβλέπουμε σε μία πρόοδο την Δευτέρα Σεπτεμβρίου. Κλείνουμε λίγο νωρίτερα από ό,τι επρόκειτο να γίνει την σημερινή μας συνεδρία. Σας υπενθυμίζω ότι αύριο η Επιτροπή μας θα συνεδριάσει στις 10.30 για να ακούσει τον κύριο Μπουζόη για την παρακολούθηση του ευρωπαϊκού δικαίου και θα υπάρξει και η παρουσίαση μιας σημαντικής μελέτης για την, τον αντίκτυπο της, της διαφήμισης στην συμπεριφορά των καταναλωτών, τον κύριο Ζουδάν και τους ε, συναδέλφους του και μια σύντομη συνεδρία στο απόγευμα για την ευρωπαϊκή τυποποίηση και τη γνωμοδότηση του κύριου Παντσέρη για το αστικό δίκαιο και το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Έτσι θα κλείσουμε λοιπόν για πριν από τις διακοπές. Οι συντονιστές φυσικά θα συνεδριάσουν από τις 9 ως τις 10.30 σε αυτή την ιδία αίθουσα. Λοιπόν, κλείνουμε για απόψε.